Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να αρχίσουμε, ακόμα και αν δεν είμαστε ακόμα αρκετά πολύ αριθμοί. Πάντως η σημαντική είναι οι παρόντες. Um, uh, αρχίσουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερησίας διάταξης, ανακοινώσει του Προέδρου και έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Προτείνω να αφαιρεθεί το 4, από την ημερήσια διάταξη και να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι το θέμα της κυρίας Κιγιόμ και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ε, ένα σχέδιο γνωμοδότησης του Προέδρου προς την Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών θα προσθεθεί ο σημείο 16α στην ημερήσια διάταξη για λόγους κατεπήγοντες. Αφορά πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και την προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων, δηλαδή τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και χρειάζεται άμεση ανταπόκριση σε αυτό. Μπορούμε να εγκρίνουμε με αυτές τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα ήθελα να σας ζητήσω επίσης την έγκρισή σας για τους εξής διορισμούς εισηγητών. Νίλ Στόρβαλτς ε, των Φιλελευθέρων για τις εξής δύο εκθέσεις. Συγχρηματοδότηση, και ποσοστό δηλαδή του Ταμείου ε, Μεταναστών, Επιστροφών και ένταξη Υπηκών Τρίτων Χωρών και το ζήτημα συγχρηματοδότησης και ποσοστό ορισμένων κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αυτό τον καιρό ε, ως προς την χρηματοοικονομική τους ε, σταθερότητα. Η ίδια πρωτοβουλία έκθεση για το πρόγραμμα τη Στοκόλμη και την εφαρμογή του εισηγητή ορίστηκε ο κύριο Λόπης Ακύλα. Ο κύριο Γιώργο Παπα-Νικολάου, συντάκτη νομοδότηση για την νομοδότηση για την απαλλαγή του οικονομικού έτου 2011. Ε, συμφωνεί η Επιτροπή με τους διορισμούς αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγκρίνεται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 27ης και 28ης Φεβρουαρίου, αλλά και της 20ης Οκτωβρίου του 2011, για κάποιο μυστήριο λόγο. Δεν έχετε σχόλια. Α, μπορείτε να φέρετε και αντιρρήσεις μέχρι αύριο το μεσημέρι, ε, το βράδυ αν κατάλαβα καλά μέχρι την αυριανή συνεδρίαση, άρα δεν πρέπει τώρα να το εγκρίνουμε αυτό το θέμα των πρακτικών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την έκθεση της κυρίας Γιγιόμ, είπαμε ότι αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, οπότε ερχόμαστε στο σημείο 5. Η ένταξη των μεταναστών του κυρίου Κλάση έκθεση. Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειε τη στην αγορά εργασία και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού τη κοινωνική ασφάλιση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και θα ήθελα καταρχάς να παρακαλέσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης να μας την παρουσιάσει και μετά να γίνει συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Κλάς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Λοιπόν, τι μας ζήτησαν εμάς ως Επιτροπή ε, Ελευθεριών. Να κάνουμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας στα κράτη-μέλη. Το κείμενο το έχετε στα χέρια σας και υποθέτω ότι οι περισσότεροι παρόντες ε, το έχουν ε, διαβάσει. Ίσως να σας εξηγήσω λίγο ε, τη φιλοσοφία της πρότασής μου. Θα ήθελα να εισάγουμε εδώ κάποια πράγματα που δεν εμφανίζονται συνήθως σε κείμενα της δικής μας Επιτροπής ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά όταν μιλούμε για τα προβλήματα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών. Καταρχάς ε, μιλώ για την προβληματική της ε, δυνατότητας απορρόφησης διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι διαφέρει πολύ η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη, τα παλαιότερα ας πούμε, στην Ένωση, που έχουν προβλήματα. Έχουμε φέρει πολλούς ανθρώπους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να τους απορροφήσουμε και να έχουν στέγη, εργασία και άλλα τινά. Καταλαβαίνετε περί ε, τίνος πρόκειται και τι εννοώ. Αν κοιτάξετε μια πόλη σαν τις Βρυξέλλες, θα καταλάβετε τι επικρατεί και ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες οι προκλήσεις για το μέλλον. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα, φέραμε κόσμο χωρίς να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε μια προοπτική για εργασία και περί αυτού πρόκειται στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει δουλειά για να φέρνουμε κόσμο και μετά να δούμε και το προφίλ τους. Γιατί συχνά τι γίνεται. Έχουμε συστήματα συνένωσης, επανένωσης οικογενειών και καμιά φορά και ε, ασύλου έρχεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, γιατί δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα σε πολλά κράτη-μέλη. Και έτσι έχουμε φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε καμία προοπτική για εργασία. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα ανεργίας, ε, κοινωνική κοινωνικής περιθωριοποίησης, γετοποίησης και πάει λέγοντας. Οπότε... Το πρόβλημα είναι οι ε, άνθρωποι με χαμηλή ειδικευση, ακόμα και ανειδίκευτοι οι ε, καινούργοι που έρχονται. Θα πρέπει να αναφέρονται και να ε, μελετάτε και το κόστος για τα κοινωνικά μας συστήματα πριν έρθουν. Επίσης, στην πρώτη συζήτηση αυτής της γνωμοδότησης το είχα ξαναπεί, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ νομίμων και παρανόμων μεταναστών. Αυτοί που έρχονται εδώ παράνομα, εντάξει, επιλογή του είναι, αλλά δεν μπορεί να περιμένουν ότι θα έχουν την ίδια μεταχείριση με κάποιον μετανάστη που φτάνει στην Ένωση νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος. Βέβαια τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν την πολιτική τους από εκεί και πέρα, αλλά κάποιος που ε, διαπιστωμένα έχει μπει παράνομα ε, στην Ένωση θα πρέπει να επιστρέφει στην πατρίδα του. Αυτά πιστεύω. Αυτή είναι η γνωμοδότηση που θα πρέπει να δώσουμε εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει το λόγο γι' αυτό. Ο κύριος Μπρόνς πρώτος και μετά θα κάνω κατάλογο. Right, um, <clears throat> as Mr. Όπως ε, είπε και ο κύριος ε, Κλάς, η γύρανση του πληθυσμού των εθνών της Ευρώπης συχνά χρησιμοποιείται ως αιτιολογία για τη μετανάστευση. Γιατί γυράσει και ο πληθυσμός, ε, φυσικά αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής και βέβαια χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ειδικά θα σας κάποια στην ηλικία μου, αλλά αλλά επειδή έχουμε και μείωση στις γεννήσεις, ε, γιατί γίνεται αυτό σε κάποιο βαθμό λόγω των εθνικών πολιτικών ε, των κρατών μελών. Πολλές φορές ε, υπάρχουν, υπάρχει ανισότητα των δύο φύλων στην, στο, στο χώρο εργασίας, ε, όμως ε, φυσικά θα έπρεπε ε, να αλλάξουν οι πολιτικές και δεν θα έπρεπε να υιοθετηθούν από τα κράτη ακραία μέτρα όπως να φέρουν μεγάλα ποσοστά ανθρώπων να τους αντικαταστήσουν ε, και αν δούμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον επαγγελματικό τομέα μπορούμε να καταρτήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ε, δεν ε, αναφέρω συχνά τους λόγους τα λόγια της Κομισιόν, αλλά στο έγγραφο του 2010 που φέρει το τίτλο Ευρώπη το 2020, σε λέει η Ευρώπη έχει πάρα πολλές δυνάμεις και μπορούμε να βασιστούμε στα ταλέντα και τη δημιουργικότητα των δικών μας ανθρώπων και η Κομισιόν έχει γράψει αληθινά λόγια. Η πολιτική της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι ε, ουσιαστικά ε, στον τρίτο κόσμο ε, να αφαιρέσει από αυτόν τον τρίτο κόσμο τους ανθρώπους που έχουν προσόντα να φέρουμε νέους μετανάστες στην Ευρώπη από τον τρίτο κόσμο για να εργαστούν εδώ σε Ευρωπαίοι. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Η κουλτούρα των ε, ε, μεταναστών ε, δεν είναι ότι θα τους δίσουμε με διαφορετικά ρούχα φέροντας τους εδώ. Υπάρχουν πιο ανεξίδηλοι πολιτισμοί και όταν έρχονται σε μεγάλο αριθμό οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη, ορισμένα τμήματα της Ευρώπης μετατρέπονται σε τρίτο κόσμο. Φυσικά οι φιλοξενούσε χώρε, οι χώρε υποδοχή θα μπορούσαν να σκεφτούν εμεί τουλάχιστον μπορούμε να αποφασίσουμε για τον αριθμό των ατόμων που δεχόμαστε. Αλλά όπω αναγνώρισε και ο συγητής στην έκθεση, για κάθε έναν ενήλικα ε, άνδρα συνήθω, τα έθνη τη Ευρώπη, τελικά πρέπει να δεκτούν και πάρα πολλού άλλου ε, και εξαρτημένα παιδιά γιατί υπάρχει και η οικογενειακή επανένωση η ε, περιγραφή που γίνεται στην έκθεση ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν αιτιολογείται η παρουσία των ανθρώπων αυτών και πολλά από τα πανεπιστήμια που λένε ότι πηγαίνουν πολλές φορές δεν υπάρχουν και μάλιστα όσοι πολλές φορές παρακολουθούν τα μαθήματα ε, συχνά παραμένουν για να εργαστούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και κάτι τελευταίο όπως ε, αναφέρεται από τον Σίτη, η, ιδέα της ελεύθερης μετακίνησης για εργασία ε, ουσιαστικά είναι παράλογη όταν έχουμε πάρα πολλούς ε, ανέργους και θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι μια τρέλα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μπρόντς. Γι' αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη φαίνεται να έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά για τα επόμενα σημεία στην ημερήσια διάταξη θα σας ζητήσω να είστε κάπως ε, πιο συνοπτικοί. Κύριε Σίκολ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει πολλά ε, σαν όσα ακούσαμε. Εγώ θα περιοριστώ ουσιαστικά σε δύο. Πρώτον, εγώ δεν θεωρώ ότι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών θα πρέπει να καταργηθεί ε, γιατί ελπίζουμε να γεννηθούν περισσότερα παιδιά. Η λύση μπορεί να βρεθεί από αλλού οι άντρες και οι γυναίκες να έχουν ενισχυμένες ευκαιρίες για να μπορούν να συνδυάζουν αρμονικά ε, το επάγγελμα με την οικογενειακή ζωή. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τον αποκλεισμό και την κετοποίηση ανθρώπων από άλλες χώρες επειδή είναι φτωχοί και ίσως όχι τόσο μορφωμένοι, αυτό το μορφωμένοι χωράει πολλή συζήτηση, ε, θέλω να πω εδώ ότι ο αποκλεισμός και η εγκαιτοποίηση συμβαίνει και στις χώρες μας απέναντι ε, σε πολίτες ε, αυτόχθονες όταν είναι φτωχοί. Δεν είναι πρόβλημα μετανάστευσης. Παρακαλώ να μην αναμειγνύουμε διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φλότρ. Για το θέμα της ε, μετανάστευσης ε, θα υπάρξει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας ε, και για τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις και πολιτιστικές διαστάσεις και τον αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση που έχουμε ενώπιόν μας ουσιαστικά παραλαμβάνει όλες τις κοινοτοπίες που ακούμε για το μεταναστευτικό ζήτημα και βασίζομαι στο έργο που μπορεί να κάνει αυτή η Επιτροπή για να τροποποιήσει αυτή τη γνωμοδότηση και επίσης ε, και ε, στο έργο της Επιτροπής Απασχόλησης που είναι η κατουσίαν αρμόδια επιτροπή και επίση πρέπει να ε, δούμε κάποια πράγματα εις βάθος. Σε αντίθεση με αυτά που συχνά λέγονται και επαναλαμβάνονται δεν είναι η πιο φτωχοί άνθρωποι που μεταναστεύουν, αλλά το αντίθετο συνήθως ε, άνθρωποι που έχουν ένα οικονομικό κεφάλαιο και ένα μορφωτικό κεφάλαιο, γιατί έχουν και κάποιους πόρους για να μπορέσουν να μεταναστεύσουν. Αυτοί έρχονται στην Ευρώπη, έτσι λοιπόν το επίπεδο της μόρφωσής τους ε, και όσο περνούν ε, τα χρόνια προσεγγίζει το επίπεδο της μόρφωσης των δικών μας πολιτών και υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στην ικανότητα των κοινωνιών μας ε, να απασχοληθούν αυτοί οι μετανάστες σε θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο της κατάρτισής τους και στις αρμοδιότητές τους. Και μεταξύ εισαγωγικών θα έλεγα εδώ υπάρχει εδώ μια απώλεια που μπορούν να κερδίσουν οι κοινωνίες υποδοχής, οι χώρες μας δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση στο ότι οι μετανάστες αυτοί, οι οποίοι είναι καλά καταρτισμένοι, τις περισσότερες φορές και δεν βρίσκουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν βάσει προσόντων στο επίπεδο των προσόντων τους. Και επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν προέρχονται συνήθως από τις πιο φτωχές χώρες, αλλά από αναπτυσσόμενες χώρες ε, και ε, ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν η γνωμοδότησή μας ε, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνει ιδέες ε, κοινότοπες και ψευδείς ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και κυρίως τη μετανάστευση για λόγους απασχόλησης. Επίσης τώρα αν γίνεται η ίδια κρισία αυτή μεταξύ της οικογενικής μετανάστευσης και της μετανάστευσης ε, για λόγους εργασίας και εξάφρησης απασχόλησης θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Γιατί καταρχήν ε, ε, το να ζει κάποιος στα πλαίσια μιας οικογένειας είναι ένας λόγος ένταξης. Έτσι λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε και για την ένταξη συνολικά και την δυνατότητα να υπάρχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και επίσης ε, το άτομο αυτό ε, να ε, μπορεί να μείνει στη χώρα του και να ασκήσει ένα επάγγελμα. Το, μισ... το ίμιση των μεταναστών είναι γυναίκες σήμερα. Έχουμε δει και τα στοιχεία του ΙΕ και του Διεθνού Γραφείου Εργασία μα λένε ότι έχουμε και γυναίκε μετανάστριε. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να δημιουργούμε κάποιε ψευδεί διακρίσει εδώ γιατί ε, πραγματικά διακυβεύονται πολλά. Και επίση η δική μα ε, γνωμοδότηση θα πρέπει να θέτει το ζήτημα τη νομιμοποίηση ανθρώπων που απασχολούνται, που εργάζονται τακτικά, κανονικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, αλλά εργάζονται με πραγματικές συμβάσεις εργασίας. Και ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε τα άτομα αυτά να μπορέσουν να νομιμοποιηθούν ε, βάσει τις συγκεκριμένε δραστηριότητες που ασκούν. Για τον αντίκτυπο αυτό υπάρχει μια μελέτη του London School of Economics, η οποία μας δείχνει ότι αν ομοποιήσουμε ε, τους 118.000 ε, ε, ανθρώπους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που θα προστίθενταν στα ταμεία του Βρετανικού κράτους. Και υπάρχουν καλά αριθμητικά στοιχεία Νομίζω ότι όταν συντάσσει κάποιο μια τέτοια γνωμοδότηση θα πρέπει να την τεκμηριώσει κιόλα. Αλλά και εγώ θα μπορούσα να δώσω στον κύριο Κλέζ μια γαλλική μελέτη που δείχνει ότι οι μετανάστε το 2010 ε, μπόρεσαν ε, να συμβάλλουν στο να έχει το γαλλικό κράτο 12 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως ε, δεν πρέπει να ε, έχουμε εδώ δηλώσεις ε, που αυξάνουν φαινόμενα λαϊκισμού, ρατσισμού. Όμως η δική μας ευθύνη ως βουλευτές είναι να ξεκινάμε από συγκεκριμένα δεδομένα που έχουν τεχμηριωθεί από τους εμπειρογνώμονες και να διατυπώνουμε προτάσεις που να στέκουν. Και το λέει και η Κομπισιόν, όποιος θέλει να το ακούσει, επαναλαμβάνει ότι η συνεισφορά των μεταναστών στην ανάπτυξη δεν μπορεί να αφιστεθεί. Δεν ε, θέλω να μιλήσω και για τη δημογραφία, γιατί μακρηγόρησα μπορούμε μόνος να προσθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Στον κατάλογο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέλστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω παρατηρήσεις για δύο θέματα που ακούσαμε εδώ στην έκθεση. Η ικανότητα ή δυνατότητα απορρόφησης. Το 1943 έγραψε ένας συγγραφέας ένα άρθρο ε, για την προετοιμασία της ε, απόβασης στην Ορμανδία. Έφτασαν οι πρώτοι Αμερικανοί και τους υποδέχτηκαν με ανοιχτέ τις αγκάλες στη Βρετανία. Μετά όμως όταν αυξήθηκαν και ήταν το 10% των ενόπλων δυνάμεων οι Αμερικανοί, οι ε, Βρετανοί τους αντιμετώπισαν με μεγάλη και αυξανόμενη αποστροφή. Και μάλιστα ήταν αμοιβαίο αυτό, the bridge and the youngs και τελικά ε, άρχισαν μεταξύ τους να συμπλέκονται κιόλας και τους χώρισαν με τρόπο αρκετά ε, αυστηρό. Και αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν κοινή γλώσσα, κοινή κουλτούρα, κοινό πολιτισμό, κοινό εργαλείο. Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης και ε, εξαρτάται αυτή από πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά ε, θα είναι ανόητο να το παραγνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο. Κάθε χώρα έχει και κάθε κοινωνία μια δυνατότητα απορρόφησης. Υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσελκύει μορφωμένους ε, αλλοδαπούς, ε, κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά είναι πώς ζουν στη χώρα. Εδώ έχουμε ε, στη χώρα μας πολίτες που δεν μπορούν να μορφωθούν ε, αρκετά ή να ε, προχωρήσουν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση για να έχουν πρόσβαση στην εργασία. Ενώ στις χώρες των μεταναστών παρατηρείται διαρροή εγκεφάλων και η χώρα καταστρέφεται. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, είναι να έχουμε μια μεταναστευτική πολιτική που δεν θα είναι απορρόφηση ε, των πιο ε, προσοντούχων ας πούμε, εργαζομένων. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια έκθεση για τη μετανάστευση. Και πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο μετανάστευση. Συγκεκριμένα, θέλουμε να πούμε οικονομική μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα σε δευτεροκλασσάτες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοκλασσάτες θεωρείται αυτό μετανάστευση και πότε νομίζετε πως θα είναι κατάλληλη η ώρα να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο διότι εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρη δικαιώματα. Εάν δούμε όμω την πραγματικότητα θα διαπιστώσουμε ότι η Ουγγαρία καθώ και πολλά άλλα από τα νέα κράτη-μέλη είναι έχουν καθεστώς δεύτερης κατηγορίας και ολόνα και περισσότεροι άνθρωποι μεταναστεύουν ως οικονομική μετανάστες, οικονομικού λόγου από τι χώρε μας στα παλαιά κρατημέλη. Και μου φαίνεται πως κανείς δεν θέλει να θίξει αυτό το ζήτημα. Μετά την δημοκρατική μετάβαση, την επωνομαζόμενη δημοκρατική μετάβαση, η βιομηχανία μας ε, ιδιωτικοποιήθηκε και εξαιτίας της ε, παγκοσμιοποίησης και της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσαμε τις αγορές μας, χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας, έμειναν άνεργοι πάρα πολλοί άνθρωποι και εκείνοι που διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους ε, ήταν γιατροί ή για παράδειγμα νοσοκόμες, αυτοί δουλεύουν, δούλευαν για 300 ευρώ το μήνα. Και οι υπάλληλοι που δούλευαν για πολυεθνικές εταιρείες και σε εργοστάσια, πολλές φορές έκαναν βάρδιες 12 ώρες χωρίς καμία νομική προστασία. Πληρώνονται περίπου 250 έως 300 ευρώ το μήνα και φυσικά πολλοί από αυτούς μεταναστεύουν μέσα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο ασχολείται με αυτού, με τη δική τους κατάσταση. Όταν μιλάμε για μετανάστευση, συμπεριλαμβάνουμε και αυτού τους ανθρώπους. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, εάν ασχολήθηκε με το φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά, όσοι μεταναστεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν δικαιώματα. Παρατηρείται φαινόμενο τράφικινγκ, το οποίο είναι, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει στον τρίτο κόσμο. Και πολύ συχνά τους παίρνουν τα διαβατήρια, δεν τους πληρώνουν, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετικά με τα κοινωνικά τους δικαιώματα, γίνεται διακίνηση γυναικών. Έχω δει για παράδειγμα γυναίκες που δεν πηγαίνουν από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις κατοχώρες στην Ουγγαρία, αλλά πολλές που πηγαίνουν από την Ουγγαρία στην Γερμανία και στις κατοχώρες. Πότε θα αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και για πόσο καιρό θα το κρύβουμε και θα το κρατάμε μυστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρφα. Πιστεύω πως το ζήτημα της ε, διακίνηση ανθρώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε ασχοληθεί πολλέ φορέ με αυτό. Δεν πιστεύω λοιπόν πώ ε, το αγνοούμε. Αλλά πράγματι αξίζει την προσοχή μα. Ο τελευταίο ομιλητή είναι ο Τζιν Μέμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την εσωτερική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την κινητικότητα του χρόνου, έχουμε το ευρωπαϊκό των πολιτών, ε, τα οποία σχεδιάστηκαν για, ακριβώς για να συζητηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρω ότι πολλά μέλη συναντήθηκαν ε, με εκπρόσωπους στα δικά τους κράτη-μέλη και ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα. Επίσης, το Κοινοβούλιο τρέχει πάρα πολλά project, ε, τα οποία βρίσκονται, για παράδειγμα, στον φετινό προϋπολογισμό και ασχολούνται, για παράδειγμα, με την πρόσβαση σε στέγαση. Και η Επιτροπή Απασχόληση ε, κάνει πολλά πράγματα για αυτό το ζήτημα και εμεί του υποστηρίζουμε. Ωστόσο, η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή τη Επιτροπή έχει να κάνει με την ένταξη. Και αυτό που ακούμε είναι μία συζήτηση για τη μετανάστευση, την οποία έχουμε διεξάγει πολλέ φορές και θα συνεχίσουμε να τη συζητάμε. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι η ένταξη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι καθήκον μας ως Επιτροπή να μιλήσουμε για αυτό. Πολλές από τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη. Για παράδειγμα, δεν συζητούμε εδώ την συμμετοχή στα κοινά, το οποίο είναι ε, μια πολύ σημαντική άποψη της ένταξης και αυτά λείπουν από την έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πιστεύω να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα ζητήματα. Και όσον αφορά τα ζητήματα για τη διαρροή εγκεφάλων, ναι, έχουμε ασχοληθεί με αυτό στο παρελθόν. Για παράδειγμα την κράτηση Ευρωπαίων πολιτών. Και επίσης το ζήτημα ότι πάρα πολλοί γιατροί, επιστήμονες δικοί μας μεταναστεύουν σε άλλες χώρες δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τους ε, ανθρώπους που έρχονται στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για λόγους εργασίας, αλλά και εκείνους που διαφεύγουν από εμάς για εργασιακούς λόγους και τη συγκράτησή τους. Τώρα όσον αφορά τα ανώτατα όρια, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε έρευνες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πιέσεις σε πολλά κράτη-μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε περιπτώσεις που κατάφεραν να ενταχθούν οι εργαζόμενοι από άλλες χώρες στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές τροπολογίες που εμείς επιθυμούμε να εισαγάγουμε και επαναλαμβάνω πως θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως μια βάση εμείς ζητήσαμε μια μελέτη από την Επιτροπή Απασχόλησης για την Εσωτερική Μετανάστευση και το πώς αυτή επηρεάζει την αγορά εργασίας. Η μελέτη δημοσιεύθηκε πέρυσι και σε αυτήν θα βρείτε πολλές πληροφορίες επιστημονικά ελεγμένες και πληροφορίες για το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού επιστρέψω στον εισηγητή, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή, κύριε Σμιτ, αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Κυρία Σμιτ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια μόνο για την ένταξη, η οποία συνδέεται άμεσα με τη μετανάστευση. Είχαμε πολλούς υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό να έχουν πλήρη δικαιώματα ένταξη για να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασία. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να το περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα και προσπαθήσαμε να το κάνουμε αρκετό καιρό πριν. Εάν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά εργασία σε ορισμένου τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε όσους βρίσκονται ήδη εδώ και όχι μόνο υπηκόους ε, άλλων ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μετανάστες που βρίσκονται ήδη εδώ και επιθυμούν να μάθουν τη γλώσσα. Πρέπει και αυτούς να τους υποστηρίξουμε. Αυτό λοιπόν αφορά την ένταξη και η ένταξη συμπεριλαμβάνει επίσης και όσους φτάνουν πρόσφατα με την έννοια ότι χρειάζονται βοήθεια για να βρουν δουλειά και να μάθουν τη γλώσσα και αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους και οι οικονομικοί μετανάστες και αυτό συνδέεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης. Και να σας υπενθυμίσω ότι φυσικά τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν τις ποσοστώσεις ε, όσων θα μπορούν να έρχονται για οικονομικούς λόγους. Και κάτι που είναι σημαντικό και είναι πρόβλημα είναι το ζήτημα που αναφέρθηκε για τη διαρροή εγκεφάλων. Ήδη υπάρχουν εδώ πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι έχουν προσόντα, αλλά τα προσόντα αυτά δεν έχουν αναγνωριστεί, οι δεξιότητε του δεν έχουν αναγνωριστεί. Επίση, ανταγωνιζόμαστε άλλες τρίτε χώρες όσον αφορά τους υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους. Και α μην ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Η ένταξη λοιπόν έχει δύο όψεις. Προσπάθειες πρέπει να γίνουν και από τις ε, κοινωνίες που δέχονται μετανάστες, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε την ένταξη σωστά πρέπει να μην ξεχνάμε γενικότερη μετανάστευση και τα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλάς, τα τελευταία σχόλια. Ναι, με ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι αυτό ε, που με ενδιαφέρει δεν είναι να έχουμε ένα συνοθήλευμα κοινών τόπων. Ήθελα να πω κάτι καινούριο. Ε, κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα ή καθόλου ή ελάχιστα. Η ικανότητα, η δυνατότητα απορρόφησης, αλλά και η διαρροή εγκεφάλων, η διαφυγή εγκεφάλων. Είναι σημαντικό αυτό και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αν θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουμε περισσότερο υπόψη την κατάσταση επιτόπου στα κράτη-μέλη. Και εκεί βλέπουμε μεγάλη ανεργία σε πολλά κράτη-μέλη. Μια ανεργία και των αλλοδαπών επίσης, όχι μόνο των ημεδαπών. Και πολύ καλύτερο θα ήταν αντί να φέρνουμε ακόμα περισσότερο κόσμο χωρίς να έχει την παραμικρή ελπίδα για εργασία, να ε, φροντίσουμε να εργαστούν όσοι βρίσκονται στην Ένωση και έτσι λύνονται περισσότερο τα προβλήματα αντί να διωγγώνονται. Με τα μεταναστευτικά ρεύματα ε, που τελικά είναι ανεξέλεγκτα. Γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα για το πόσο κοστίζει η μεταναστευτική πολιτική, ποιο είναι το καθεστώς ε, και το καθαρό κόστος ε, μετά από δεκαετίες ε, πολιτικής στα κράτη-μέλη. Εγώ είδα μια μελέτη από την Ολλανδία, από ένα γραφείο μελετών του Νάιφερ. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να το ζητήσετε και να σας τη δώσω. Και η μελέτη αυτή ε, ε, δεν επικρίθηκε από κανέναν επί της ουσίας, ε, δεν γνώρισε αντιδράσεις από πολιτικούς που είπαν ότι κοιτάξτε τι, αυτά που λέει αυτή η μελέτη δεν ισχύουν, ο υπολογισμός, η μέθοδος δεν ισχύει. Δεν έχω ακούσει τίποτα, απλώς εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είναι πολύ μικρή η διαφάνεια στα κράτη-μέλη ε, και ε, η ε, κυβέρνηση δεν δίνει τα στοιχεία που χρειάζεται κανείς για να τα υπολογίσει. Πόσο μας κοστίζει η μεταναστευτική πολιτική τελικά και ποια είναι η ανάλυση κόστους ωφέλειας. Γιατί εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι Βεβαίω και μας ωφελεί η μετανάστευση, αλλά δεν μπορούμε και να τα υπολογίσουμε. Τι γίνεται όταν έχουμε μαζική ανεργία, τι ε, γίνεται όταν δεν εντάσσονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε μόνο το δικαίωμα ως κοινοβούλιο, αλλά και το καθήκον να καθίσουμε να σκεφτούμε ε, πώς θα αλλάξουμε τακτική, ρότα, πορεία, ε, να έχουμε μια εναλλακτική πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ε, βέβαια πιο αυστηρή πολιτική με λιγότερη μετανάστευση, αλλά πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σημαίνουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας, αλλά τους δίνουμε και μια προοπτική, μια ελπίδα για ένταξη μέσω της εργασίας. Και πολύ συχνά, δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς είμαστε ωραίοι για τις μεγάλες ιδέες και τις μεγάλες αρχές και ανοίγουμε τις θύρες και μετά επιτόπου έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και προχωρούμε στο σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο νέων προτάσεων για εξυγχρονισμό το, της συγχρηματοδότησης στα ταμεία προσφύγων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξη Υπηκών Τρίτων Χωρών να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότηση κατά 20%, 20% για τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, η Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία είναι οι έξι χώρες. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις και μετά στην Κυπριακή Προεδρία για να σχολιάσει την κατάσταση των πραγμάτων στο Συμβούλιο και μετά στον εισηγητή μας τον κύριο Τόρβας αν συμφωνεί ο εισηγητής και μετά θα γίνει συζήτηση μπορώ ήδη να σας ενημερώσω ότι έχουμε κάποια χρονική πίεση. για να μπορούν να ισχύσουν για τα προγράμματα του 2011 αυτές οι αλλαγές και προτείνουμε το εξής προθεσμία κατάθεσης ε, του σχεδίου έκθεση, στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα 26 Νοεμβρίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 29 Νοεμβρίου, ψήφιση στην Επιτροπή μα 17 ή 18 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια αρχέ του 2013. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Σαβαρή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος και σύντομα στην παρουσίασή μου, καθώς πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα. Καταρχήν, όπως υπενθυμίσατε και εσείς, η πρότασή μας αποτελείται από δύο προτάσεις. Η μία αφορά το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα και άλλη που αφορά το Ταμείο ε, για την Επιστροφή, το Ταμείο των Προσφύγων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξη Υπηκών Χωρών, γιατί έχουμε δύο διαφορετικέ νομικέ βάσει. Οι δύο αποφάσει είναι σχεδόν ταυτόσιμε. Δηλαδή είναι το διατακτικό το ίδιο και έχουμε ακριβώ του ίδιου τρόπου παρουσίαση. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν διαφορέ επίπεδο περιεχομένου Αυτές οι δύο αποφάσεις ε, απλώς συνδέονται με διαφορετικές νομικές βάσεις. Ποιος είναι ο μηχανισμός λοιπόν που προτείνεται σε αυτές τις δύο αποφάσεις. Θα το γνωρίζετε ίσως, ε, έχουμε ένα σύστημα ετήσιου προγράμματος για τα ταμεία, δηλαδή η Κομισιόν κάθε χρόνο αποφαίνεται επί ενός προγράμματος που καταρτίζουν τα κράτη-μέλη με περίοδο πλεξιμότητας που διαρκεί 2,5 έτη και που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν δράσεις κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών. Για ένα ετήσιο πρόγραμμα 2010 τα κράτη-μέλη λαμβάνουν ε, μια εκταμίευση που θα του επιτρέπει να χρηματοδοτήσουν δράσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Επομένως, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουμε δύο συντελεστές χρηματοδότηση, ένα κανονικό συντελεστή του 50% και ένα πρόσθετο συντελεστή του 75%. Εδώ μιλάμε για ε, δράσεις που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων, την ένταξη κτλ. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε και ένα ποσοστό 75% που ισχύει συστηματικά για όλες τις χώρες ε, που λαμβάνουν κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Η δική μας πρόταση επιτρέπει, θέλει να επιτρέψει σε ορισμένα κράτη-μέλη που βιώνουν δυσκολίες σε οικονομικό επίπεδο να αυξήσουν κατά 20 μονάδες ε, αυτό το ποσοστό. Δηλαδή για ένα κανονικό ποσοστό 50% θα μπορούσαμε να έχουμε αύξηση στο ποσοστό της χρηματοδότησης στο 70% και για το 75% θα μπορούσαμε να φτάσουμε ε, στο 95% ε, ή θα μπορούσαμε να μιλάμε λοιπόν για χρηματοδότηση από το 75-75% για όλε τι δράσει των χωρών αυτών. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια για να μπορεί να υποφεληθεί κάποιο από το μηχανισμό αυτό. Δεν ήμασταν πρωτότυποι στην πρότασή μα, γιατί ακολουθήσαμε ακριβώ την προτείνεται στο πλαίσιο των διαφορετικών ταμείων και των ε, γεωργικών ταμείων και του Ταμείου Ελίας. Ε, αυτή η απόφαση ήδη υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Τα κριτήρια λοιπόν είναι ακριβώς τα ίδια, ανοίγει δυνατότητα στα κράτη-μέλη που ε, έχουν λάβει χρηματοοικονομική βοήθεια, τον κατάλογο το βλέπετε στην απόφαση. Πρόκειται ουσιαστικά για πέντε κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, αλλά ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε να διευρυνθεί. Ποιος είναι ο αντίκτυπος χρηματοοικονομικό, χρηματοοικονομικός, ο αντίκτυπος ε, για την εκταμίευση, για τα κονδύλια που έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη, είναι μηδενικό. Ε, δηλαδή, επιτρέπουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη που βιώνουν ε, δυσκολίες σε επίπεδο προπολογισμού να συνεισφέρουν λιγότερο από το εθνικό κονδύλι. Έτσι λοιπόν, εκεί όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν 50%, σήμερα μόνο 30% θα πρέπει να συνεισφέρουν και στην περίπτωση που θα πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά 25% ε, σήμερα θα είναι 5%. Να σας εξηγήσω και ένα τεχνικό στοιχείο, όπως επενθύμησε και η κυρία Πρόεδρος, μας πιέζει ο χρόνος για την απόφαση αυτή αν θέλουμε αυτή η απόφαση να μπορεί να εφαρμοστεί στα προγράμματα του 2011 που τρέχουν σήμερα, είναι υποεκτέλεση, θα πρέπει αυτή η απόφαση, αυτές οι αποφάσεις να θετηθούν πριν το Μάρτιο του 2013. Γιατί? Γιατί για να εφαρμόσουμε αυτό το νέο συντελεστή χρηματοδότηση, τα κράτη-μέλη πρέπει να θεωρήσουν τα αιτήσια προγραμματά του. Για να γίνει αναθεώρηση των αιτήσιων προγραμμάτων, τα κράτη-μέλη Σύμφωνα με τον κανονισμό των ταμείων θα πρέπει αυτό να γίνει τρει μήνε πριν από την περίοδο επιλοξιμότητα. Έτσι λοιπόν και τα προγράμματα του 2011 θα πρέπει οπωσδήποτε τα προγράμματα του 2011 να θεωρηθούν πριν ε, τα τέλη Μαρτίου 2013. Διαφορετικά, αυτός ο νέος μηχανισμός δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στα προγράμματα του 2011, αλλά μόνο το πρόγραμμα 2012-2013. Φαίνονται κάπως τεχνικά όλα αυτά, αλλά για ορισμένα κρατημέλη θα είναι πολύ σημαντική η διαφορά, κυρίως όταν μιλάμε για κρατη που γνωρίζουν σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες και που θα μπορούσαν έτσι να βελτιώσουν την απορρόφηση των ταμείων αυτών χάρη στο μηχανισμό αυτό και ήδη από τα προγράμματα του 2011. Ξεκινώντας με τα προγράμματα του 2011, πιστεύω να μην ξέχασα τίποτα. Για να συνοψίσω, πρόκειται για ένα απλό μηχανισμό που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη που βιώνουν χρηματοοικονομικέ δυσκολίε και δυσκολίες επίπεδο προπολογισμού, δημοσιονομικέ δυσκολίε να βελτιώσουν το επίπεδο απορρόφησης ε, των ταμείων Solid και να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα και δράσεις πολύ σημαντικά στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σεβέρη. Υπάρχει εδώ κάποιος ε, εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας. Συγγνώμη, δεν ξέρω το όνομά σας. you very much, Madam um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανταργυροπούλου λέγομαι, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου. Πολύ σύντομα, να προσθέσω σε αυτά που είπε η Κομισιόν. Οι δύο προτάσεις που έχουμε τώρα επιτάπητος είναι πολύ σημαντικές και φυσικά αποτελούν ε, μέρος της γενικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και τις ε, συνέπειες που έχει αυτή για τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να πω ότι η χρηματοοικονομική κρίση ήδη έχει πιέσει πάρα πολύ τους προπολογισμού των κρατών μελών και στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή των προγραμμάτων υπό τον Ταμείο Solid ήταν πολύ δύσκολη. Και ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο και πολύ συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ιδίω για αυτά που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και τι συνεπιέ τη. Και στο πλαίσιο αυτό έχουν λάβει χρηματοοικονομική βοήθεια, δυνάμει ενό από τους μηχανισμούς που αναφέρεται στην πρόταση. Η Προεδρία ήδη συζήτησε τις δύο προτάσεις ε, στο Συμβούλιο ΔΕΗ, σε επίπεδο συμβούλων και η γενική αίσθηση ήταν ότι ήταν αποδεκτές και οι δύο προτάσεις από το κράτη-μέλη. Όπως ε, είπε και η Κομισιόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δύο προτάσεις να εφαρμοστούν πριν από το Μάρτιο του 2013, για τους λόγους που ήδη εξηγήθηκαν με σαφήνεια από την Κομισιόν. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνα τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίε να είναι σε θέση να υποφεληθούν, να μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτέ τι δύο προτάσει για το έτος 2011 και για το 2011. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καρποφόρη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα για πάρα πολλού φακέλου. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε στο δύο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και φτάνουμε στον κύριο Τόβαλ, στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν και την Προεδρία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε. Άκουσα τα όσα υπόθηκαν από τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της Προεδρίας ε, και από την ε, Αγαπητή Πρόεδρο, συμφωνώ. Επομένως, ε, κατανοούμε ότι πιέζει ο χρόνος, ε, κατανοούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε βαρετές δηλώσεις για αυτό το πάρα πολύ τεχνικό ζήτημα. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δεν έχουν αξιολογηθεί άμεσα σε σχέση με τα όσα επικομισιώνει η Προεδρία. Πιστεύουμε ότι μία επιχείρηση στα σύνορα μπορεί να είναι αντικείμενο διαχείρισης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και δεν είμαστε πεπισμένοι ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ καλά οργανωμένα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση σύνορων. Εγώ έχω δει πάρα πολλά σύνορα δημοσιογράφο. Το χειρότερο ήταν το χειρότερο παράδειγμα, ήταν το ρωσικό παράδειγμα και είχαμε οκτώ υπηρεσίε ε, που σαμπόταραν η μία την άλλη. Και έχω το συνέστημα, έχω την αίσθηση μερικές φορέ, ότι δεν ξέρουν κάποιοι πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια υπηρεσία και όταν μιλάμε για αποδοτικά, πολλές φορές ε, μιλάμε με αρνητικό τρόπο για την αποδοτικότητα στα ε, σύνορα. Τη δεκαετία του 80 είχαμε... Ε, είχα, ε, συνάντησα έναν αστυνομικό και με ρώτησε «Έχετε όπλα» Και μπορώ να σα πω ότι μπορεί να ήταν αποδοτική η επαγγελματική ερώτηση, αλλά δεν τέθηκε με τον σωστό τρόπο. Έτσι λοιπόν, αν η Κομισιόν μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία σε σχέση με το πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των συνόρων θα το εκτιμούσαμε, γιατί έχουμε αυτό το πολυετή στρατηγικά προγράμματα, τον πολυετή στρατηγικό προγραμματισμό, Και ε, πιστεύω ότι μπορείτε να έχετε κάποια ιδέα σε σχέση με την αποδοτικότητα και με τον συνόρων και πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Κατανοούμε ότι πιέζει ο χρόνος και προσπαθούμε να είμαστε ήδη από αυτή την εβδομάδα αποτελεσματικοί. Πιθανότητα θα έχουμε μια πρώτη εκδοχή του κειμένου την Τετάρτη και όλοι όσοι ενδιαφέρονται είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν σχόλια. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο ότι οι αρχές στα σύνορα δεν φημίζονται για το χιούμορ τους. Κύριε Τριανταφυλλίδη και μετά ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. προσωπία αυτής της Επιτροπής επίσης επέστρεψε από την Ελλάδα. Και είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι από τα ταμεία αυτά. Και η πρώτη μου αντίδραση σε σχέση με τα στοιχεία που ακούσαμε από 50, 70 ή 75 σε 95% είναι καλό ο συντελεστής. Αλλά πόθεν τα χρήματα, πώς επηρεάζει αυτό τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν τα κονδύλια, υπάρχουν τα λεφτά. Και αν υπάρχουν, από πού προέρχονται, από οικονομίες που κάναμε, διότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποίησαν σωστά αυτά τα ταμεία. Θα ήθελα παρακαλώ κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Yes, um, <clears throat> I'd like to... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς πού βρίσκονται τα χρήματα για αυτά το ταμείο. Οι παράνομοι ή μη νόμιμοι μετανάστες υπόθηκε ότι δεν κρατούνται για πολύ καιρό και δεν επιστρέφονται δια της βίας στη χώρα προελευσής τους. Και τους ρώτησα με ευγενικό τρόπο να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά καθώς καταλαβαίνω δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πού θα, δαπανηθεί, πού θα δαπανηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Επιστροφής. Μετά, το Ταμείο Επιστροφής είναι ένα από τα τέσσερα ταμεία τα οποία στο παρελθόν ε, έχουν μετακινήσει κονδύλια από το ένα ταμείο στο άλλο και αναρωτιέμαι ποια είναι η στάση και η πραγματική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετέχουν. Γιάννη Μούλτερ. Ε, ναι, θα ήθελα να πω ότι είναι αναπόφευκτο να δεχτούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνει κάτι, διότι αυτές οι χώρες δεν είναι σε θέση να πληρώνουν τις εισφορές τους. Υπάρχουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες και θα είναι προ όφελο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική για να μην υπάρχουν κίνητρα σε ορισμένα κράτη-μέλη για αίτηση συγχρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει να λάβει το λόγο τότε, κύριε Τόρβαλτς, τελευταία σας σχόλια. Μάλιστα, νομίζω πως δεν έχω πολλά να πω, εκτός ίσως από το ότι θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα που θίχτηκε από τους προλήσατες. Ναι, ίσως θα θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Μπρόντς ή η Επιτροπή θα ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση του κύριου Μπρόντς. Διότι είμαι σίγουρη πως έχουν τις πληροφορίες και τους αριθμούς που θα θέλετε να μάθετε. Η Επιτροπή θα ήθελε να απαντήσει. Κυρία Σεβέρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τις τρεις ερωτήσεις που έγιναν. Ερώτηση πρώτη. Ε, του Η απάντηση συνδέεται με την αξιολόγηση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ταμείο. Ε, αυτό τον καιρό δίνουμε στα κράτη-μέλη χρήματα σε αιτήσια βάση και βάση προγράμματος ετησίου. Υπάρχουν πολλά αιτήσια προγράμματα που εφαρμόζονται ήδη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε αρχίσει μια πρώτη αξιολόγηση, ένα απολογισμό στη μέση της περίοδου. Είναι ένα πολύ μακροσκελές ερωτηματολόγιο αυτό που έχουμε στείλει στα κράτη-μέλη για να αξιολογηθούν τα πρώτα αποτελέσματα των πρώτων προγραμμάτων 2007, 2008, 2009, 2010 και τα αποτελέσματα θα έλθουν στα τέλη του έτους. Θα τα αναλύσουμε και μετά θα κάνουμε έκθεση που θα ε, σας ε, απευθυνθεί και θα συζητηθεί φαντάζομαι και στο φόρουμ αυτό. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Προς το παρόν είναι γεγονός ότι ως βάση εργασίας έχουμε μόνο τις δράσεις των προγραμμάτων αυτών των ετησίων, επαναλαμβάνω. Οπότε ε, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τον πρώτο απολογισμό των δράσεων που υλοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο. Για τη δεύτερη ερώτηση, από πού βρίσκουμε τα χρήματα. Όπως σας εξήγησα στην αρχή, υπάρχουν τα χρήματα, διότι είτε για το 2011 ε, που έχουν ήδη δοθεί τα κονδυλία για το 2012 που εγκρίνονται τώρα τα προγράμματα ή τα περισσότερα έχουν ήδη εγκριθεί για το 2013 ε, έχει οριστεί το ποσό τα κράτη-μέλη γνωρίζουν από τώρα το ποσό που τους αναλογεί για το 2013 και προετοιμάζουν τα προγράμματά τους που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 η πρότασή μας λοιπόν δεν αλλάζει τίποτα στα αριθμητικά στοιχεία αν είχε 100 ας πούμε ε, ένα κράτος μέλος, το 100 αυτό δεν αλλάζει. Αλλά ε, από εκεί που έπρεπε να χρηματοδοτεί από τα 100 τα 50, τώρα θα χρηματοδοτεί μόνο τα 30 από τον εθνικό του προπολογισμό. Δηλαδή το, η συγχρηματοδότηση του κράτους μειώνεται. Σε σχέση με το παρελθόν, πριν εγκριθεί αυτός ο μηχανισμός. Ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, των πόρων από το Ταμείο Επιστροφής. Έγινε μια πρώτη ανάλυση βάσει πάλι των ετησίων προγραμμάτων ε, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Επιστροφής και αυτή κατέδειξε ότι τρεις είναι οι βασικές ε, χρήσεις για το Ταμείο Επιστροφής. Έχουμε τις δράσεις τις ίδιες επαναπατρισμού ή επιστροφής είτε είναι επαναπροώθηση αναγκαστική είτε θελούσια αποχώρηση και βλέπουμε ότι οι θελούσιες αποχωρήσεις έχουν αυξηθεί και έχουν μειωθεί λίγο οι αναγκαστικές επαναπροωθήσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων και υπάρχει και ένας αριθμός δράσεων που αναφέρονται στην ενημέρωση, ε, στην κατάρτιση για θέματα σχετικά με επιστροφές για εκείνους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία αν θέλουν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν και ε, αλλαγή ε, των πρακτικών επίσης μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων αρχών και ακόμα δράσεις για τη χρηματοδότηση της ανακαίνησης κέντρων κράτησης, εργασίες δηλαδή, αναμονή εκείνων που περιμένουν να επαναπατριστούν. Αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Επιστροφής και εγγράφονται σε ένα πλαίσιο που ε, ορίζεται από την οδηγία την ε, σχετική για την επιστροφή. Και πάντα χρηματοδότηση γίνεται σε πλήρη σεβασμό του πλαισίου της οδηγίας. Αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 4.30 σε μισή ώρα. Απουσιάζει και η συγγήτρια. Οπότε τι να κάνουμε. Διάλειμμα. Μέχρι τις 4.30 προτείνω. Συμφωνείτε. Ραντεβού στις 4.30.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 Να ξαναρχίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπω ότι έχει φτάσει και η συγγήτρια. περάσουμε στο συνολικό τη ημερήσια διάταξη κατάσταση των συνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ναταλή Γκρίσπερ και είναι η συγγήτρια στις 18 Οκτωβρίου η διάσκεψη των Προεδρών επέτρεψε ανάθεση στη ΛΥΜΠΕ να καταρτήσει δυνάμει του κανόνα 48, μια έκθεση πρωτοβουλία. Σήμερα θα ακούσουμε την εισηγήτρια και κατόπιν ε, θα δώσουμε ε, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία στην διάμεση επισκόπηση τη εφαρμογή του σχέδιου δράση για του συνόδου ανηλίκου που δημοσιεύτηκε ε, στι 28 Σεπτεμβρίου και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσουμε του εκπροσώπου του γραφείου ε, τη ΥΠΑ των Εθνών για του πρόσφυγε και από τη UNICEF που θα μα παρουσιάσουν τη μελέτη του για τη δικαστική εφαρμογή του άρθρου 3 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρίσπερκ και κατόπιν στους υπόλοιπους ομιλητές και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε περίπου μία ώρα για τη συζήτηση αυτή στη διάθεσή μας. Εσείς λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να μην μακρηγορήσετε. Παρακαλώ, κυρία Κρίσπερκ, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που διορίστηκα συγχύτρια για ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα κεφαλαιόδες και ουσιαστικό ζήτημα για όλα τα μέλη της Επιτροπής Λίμπης και αφορά την κατάσταση των ασυνόδευτων ενηλίκων ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα ήθελα ήδη να ευχηθώ το επόμενο εξάμεινο εργασιών να μας επιτρέψει να εκπονήσουμε ένα ποιοτικό έγγραφο και ένα έγγραφο που θα απαντά στις θεμελιώδεις και ολοκληρών και αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών αυτών που βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση παντού, όχι μόνο στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και στο ιστορικό των κρατών μελών. Πριν ε, να περάσουμε σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα ήθελα να καταλήξουμε όλοι μαζί στο να δημιουργήσουμε ένα νομικό εργαλείο, ένα νομικό μέσο συνεκτικό, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία δράσης, χρήσιμα για τα κράτη-μέλη και που θα επιτρέπει να ομαδοποιείται τα ειδικά χαρακτηριστικά των ασυνόδευτων υλίκων ε, στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω το γενικό πλαίσιο της έκθεσης αυτής, να υπενθυμίσω όχι δε ψηλά αριθμητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας ε, ή ε, τα στοιχεία που έχουμε κυρίως σε ό,τι αφορά τους ετούντες άσυλο, αλλά θα ήθελα σε γενικές γραμμές να υπενθυμίσω ότι το ίμιση των εκτοπισμένων ε, στον κόσμο και των προσφύγων στον κόσμο είναι παιδιά. Και κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά φτάνουν στην Ευρώπη, κάποια με την οικογένειά τους και πολλά χωρίς βρει. Ασυνόδευτα παιδιά λοιπόν εγκαταλείπουν αυτά τα παιδιά τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τη βία, τις βιοπραξίε, τις διώξεις, τη παραβίαση των θεμελιωδών τους ε, δικαιωμάτων τους ε, ή φυσικές καταστροφές. Τα παιδιά αυτά Επίσης, ε, δυστυχώς μερικές φορές είναι θύματα εμπορίας, ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ε, και αντικείμενο του οργανωμένου εγκλήματος που καταπολεμούμε με πάρα πολλά νομοθετικά μέσα και ξέρετε ότι πολύ συχνά δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα μέσω των κειμένων μας και εγώ θέλω να επαναλάβω ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα, αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων και επίσης όταν φτάνουν σε μια ξένη χώρα είναι ακόμη πιο ευάλωτα γιατί υπάρχει ένας διαφορετικός πολιτισμός, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη γλώσσα και δεν είναι μαζί με την οικογένειά τους, με τους γονείς τους, με τον κεδεμόνα τους ή με οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε ε, άνθρωπο που να μπορεί να τους βοηθήσει. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όλα έχουν υπογράψει εδώ και πολύ καιρό πολύ άριθμα διεθνή νομοθετήματα της ε, Σύμβαση, τη Σύμβαση των ΗΠΑ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ. Επίσης, τη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιωμάτων, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, της Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διορθώνω μιλήτρια και αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, συνόδου των ανηλίκων, αυτών των παιδιών, ε, δεν γίνονται σεβαστά σε καμία περίπτωση, Δυστυχώ Και αυτό ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είτε να ασυνόδευτα αυτά τα παιδιά, είτε όχι, ε, τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλε. Δυσκολίε σε όλα τα στάδια τη μεταναστευτική διαδικασία Του συμπεριφέρονται ως λαθρομετανάστες, ενήλικου και τα ειδικά δικαιώματα τους και οι ανάγκες τους ε, δεν λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. Δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου, μπορεί να τεθούν υποκράτηση σε ε, τέτοια κέντρα φιλοξενίας με ενηλίκους, με συνθήκες που δεν επιτρέπονται για παιδιά, παράδειξη συνθήκες για παιδιά, χωρίς να έχουν ε, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και σε βασικές ε, υπηρεσίες και μπορεί να επαναπατριστούν χωρίς να γίνει αξιολόγηση των αναγκών τους για προστασία, μπορεί να μην λαμβάνουν ε, πληροφορία σε γλώσσα που να καταλαβαίνουν, ε, δεν έχουν το δικαίωμα να εκφραστούν κατά τη διάρκεια διαδικασίας και δεν έχουν πάντοτε νομική βοήθεια δύο γρήγορα παραδείγματα που μας ε, δείχνουν την αγκαιότητα να εγγυθούμε ελάχιστα πρότυπα για αυτούς τους ενηλίκους ε, έναντι των σημερινών ε, τάσεων και του μηχανισμού κατά των δαστών που αναπτύσσεται σε πολυ άριθμα κράτη-μέλη. Καταρχήν, ε, θα αναφερθώ σε κάτι που αφορά τη χώρα μου. Η Γαλλία δεν είναι πάντοτε παραδειγματική και πάλι καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αρχή του ε, στην απόφαση Πόποφ κατά της Γαλλίας για παραβίαση του άρθρου 3, για ε, μεταχείριση απάνθρωπη. Ε, και καταδικάστηκε η Γαλλία επειδή έθεσε υποκράτηση ε, δύο παιδιά, ένα παιδί δύο μηνών και ένα κορτσάκι τριών ετών για δύο μήνες ε, σε κλειστό κέντρο κράτησης. Υπήρξε λοιπόν παραβίαση του άρθρου 3 και το δικαστήριο απεφάνθη ότι οι συνθήκες κράτησης δεν επέτρεπαν την κανονική ανάπτυξη των παιδιών και στην περίπτωση αυτή ήταν και συνοδευόμενα τα παιδιά. Δεύτερο παράδειγμα εντάχει. Αλλά μας δείχνει πολλά. Έχουμε την απόφαση Ράιμι κατά της Ελλάδας, όπου το δικαστήριο του Στρασβούργου καταδίκασε την Ελλάδα το 2011 και άλλη παραβίαση του άρθρου 3. Ένας Αφγανός 15 ετών συνελήφθη από την αστυνομία στη Λέσβο και τέθηκε υποκράτηση στο κέντρο της Παγανής και αναφέρω εδώ την απόφαση 200 άτομα ε, μοιράζονται δύο τολέτες, κοιμούνται στο πάτωμα δεν υπάρχει ε, ουσιαστικά αέρας, ε, υπάρχουν στρώματα ε, βρεγμένα στο έδαφος και το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν γίνει, υπάρχει σεβασμός στην αξιόπινη της σε αυτές τις συνθήκες και δεν μπορεί να υπάρξει κράτηση από τι συνθήκε αυτές. Έτσι λοιπόν, ε, σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε και του συνομιλητέ μας. Ε, έχουμε ε, πολλές υποθέσεις, δυσεπίλητε. αφορούν την πρόσβαση στην επικράτεια, το δικαίωμα διαμονής, το πρόβλημα της επαναπροώθησης, στα σύνορα, το πρόβλημα της απομάκρυνσης από την επικράτεια, το θέμα της ε, ε φιλοξενίας συγκράτησης αν θέλετε, το θέμα της ένταξης, ε, της ε, συνθήκες, της άδεια παραμονής, το πρόβλημα που συνδέεται με την οικογενειακή επανένωση και την υποκρέωση τα κράτη να αναζητήσουν τους γονείς των συνοδευτών ενηλίκων. Βέβαια, το πρόβλημα της αξιολόγησης της ηλικία, ε, της νομικής εκπροσώπησης, της νομικής βοήθειας, ε, της πρόσβασης της προστασίας, της προστασικής κοινωνικής υπηρεσίας, της αναζήτηση σε όπως αποκαλεί η νομολογία του του συμφέροντος ε, του παιδιού και αυτό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αυτά όλα θα παρουσιάσει, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει αυτή η έκθεση πρωτοβουλία ε, το του να πιο συγκεκριμένο τρόπο. Και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα μέτρα, να προκύψουν από αυτή την έκθεση συγκεκριμένα μέτρα. Οι εργασίε μα ε, ελπίζω ε, ότι στους επόμενους μήνες θα απαντήσουν σε όλα αυτά τα πολύπλοκά ζητήματα. Κατανοούμε ότι η κατάσταση αυτών των παιδιών που έρχονται στην Ευρώπη είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί επιγόντως και δεν ε, ε, είναι ένα θέμα που μπορούμε να το παραγωνίσουμε καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και πολύ καιρό το Κοινοβουλίο ζητά νομοθεσία, ζητά ελάχιστα πρότυπα στον τομέα αυτό κοινοτικά νομοθετήματα υπάρχουν και πολλοί άριθμα και γίνεται αριθμός, ε, γίνεται με συγχωρείτε αναφορά στο Συνόδο της Ανηλίκου, αλλά χρειαζόμαστε ένα καθολικό συνεκτικό νομοθετήμα για το θέμα αυτό και συγκεκριμένο. Και είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε μια νομοθεσία, ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε συνολικά την κατάσταση των ανηλίκων. Για να ολοκληρώσω, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εγώ θα ήθελα, και ελπίζω να συμφωνούν συνάδελφοι, στη σύνταξη του κειμένου αυτού να γίνει από την, ε, από την οπτική των παιδιών. Δηλαδή όχι μόνο από την σκοπιά του δικαιώματος ασύλου, αλλά θέλαμε να έχουμε μία κάλυψη του συνολικού φαινομένου της μετανάστευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, παρουσιάσουμε πώς θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τα ιδεώδη της ασφάλειας και της ελευθερίας που αποτελούν το θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Συγχύτρια. Δεν θέλω να σας διακόψω για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά κοιτάζω και το ρολόι και θα παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές πραγματικά να τηρήσουν ε, το δεκάλεπτο ούτε και λιγότερο παρακαλώ. 7,5 έκαστος. Αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Αν θέλετε να δευτερολογήσετε κιόλας να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Θα χρειαστεί πραγματικά να είναι όσο πιο σύντομη η παρέμβασή σας. Ο κύριος Σμίτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε, ιδιαίτερα στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, ε, αυτό το θέμα με μεγάλη άφηξη ασυνόδευτων ανηλίκων. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνει κάτι και προτάθηκε και ένα πρόγραμμα δράσης, ε, συμφώνησε το Συμβούλιο. Θα πω δύο λόγια γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Σεπτεμβρίου ε, έφερε την ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή και περιγράφει τα όσα έγιναν και σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και τι έχουν κάνει οι οργανισμοί και της Ένωσης και των κρατών μελών ε, διεθνείς οργανισμοί και η κοινωνία των πολιτών επίσης ενημερώθηκαν. Ποια ήταν τα κύρια ευρήματα. Καταρχάς, αυτό που είπε η κυρία Γκρισπέκ, το φαινόμενο δεν είναι προσωρινό, είναι μάλλον μόνιμο ε, ε, και στο μέλλον θα έχουμε μεταναστευτικά ρεύματα, γι' αυτό χρειάζεται μια κοινή ε, προσέγγιση όπως ορίζει και το πρόγραμμα δράσης αυτό επιβεβαιώνεται. Για ποιο λόγο μεταναστεύουν ασυνόδευτοι οι ανήλικοι. Είναι περίπλοκοι, αναφέρθηκαν ορισμένοι λόγοι και ανεξάρτητα από τους λόγους, θα πρέπει οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να θεωρούνται πρώτα παιδιά και μετά μετανάστες. Ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι έχει γίνει τώρα ε, κατά τη διετία αυτή. Το πρόγραμμα δράσης ενίσχυσε ε, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ διαφόρων οργανισμών ε, μαθαίνουν τα κράτη-μέλη από τις επιτυχίες ε, τα, ε, αλλά και από, από τις λιγότερο επιτυχείς καταστάσεις ή τις αδυναμίες. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διακίνηση ανθρώπων ή μη ασφαλής αποχώρησή τους και θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται και οι συνοριοφύλακες ε, και των χωρών όταν φτάνουν στα σύνορα συνόδευτοι ανήλικοι. Έχουν γίνει προγράμματα κατάρτισης ε, χάρη στις προσπάθειες της Frontex και ε, του ΕΑΣΟ για να καταρτιστούν οι υπάλληλοι σε αυτά τα θέματα. Επίσης χρηματοδόθηκαν προγράμματα για την συνειδητοποίηση, για ειδική κατάρτιση, για να αναγνωρίζουν οι ενεχόμενοι υπάλληλοι καταστάσεις κινδύνου. Συστήθηκε και μια ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, δύο ε, αντίστοιχε συνεδριάσει έγιναν σε δύο χρόνια για την φύλαξη των ανηλίκων αυτών και για την αναζήτηση των οικογενειών Ανταλλαγή λοιπόν πρακτικών και χρηματοδότηση χρειάζεται για ε, τη διάδοση της πραγματογνωμοσύνης. Το πρόγραμμα δράσης όμως δεν αφορά μόνο την ανταλλαγή εμπειριών και τις κοινέ εμπειρίες, ε, αλλά και την εφαρμογή της νομοθεσίας και της υφισταμένης κείμενης, αλλά και της εκπόνησης ε, νέας γενοτικής νομοθεσίας για το άσυλο, για τη διακίνηση ανθρώπων, το τράφικινγκ δηλαδή. Και ε, όλα αυτά ε, προς το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και ε, γενικότερα των ασυνόδευτων αλήκων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην οδηγία της Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και της ε, ταυτοποίησης των θυμάτων ε, πέρυσι ετέθη σε ισχύ αυτή και μέχρι την 6η Απριλίου του 2013 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να την έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία. Ορίζεται εκεί σαφώς ε, τι ισχύει και τι πρέπει κανείς να κάνει για να προστατεύει ασυνόδευτους ανηλίκους. Όπως ορίζει το πρόγραμμα δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να τροποποιήσει την νομοθεσία για το άσυλο. Αυτό σημαίνει βελτίωση και της πολιτικής απέναντι σε ασυνόδευτους ανηλίκους, γιατί είναι ευάλωτοι, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία ασύλου και θα πρέπει αυτό να την υπόψη. Πολιτική συμφωνία ε, για την οδηγία για την υποδοχή και τον κανονισμό του Δουβλίνου με αυξημένες εγγυήσεις για ε, τους ασυνόδευτους ανηλίκους που αιτούν άσυλο. Δηλαδή θα πρέπει πάντα να ορίζεται ένας νομικός αντιπρόσωπος που να έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ανηλίκων. Και υπάρχει και ένα νομικό μέσο που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει τα κράτη-μέλη αλλά αναμένεται να συμφωνήσουν μέχρι τα τέλη του έτους και αφορά την οδηγία για το άσυλο αυτό ε, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό να εξαιρούνται οι ε, ανήλικοι από κάποιες διαδικασίες στα σύνορα, ας πούμε η κράτηση των ετούντων που δεν προσφέρονται για ανηλίκους. Ε, ελπίζουμε να συμφωνηθεί η οδηγία αυτή με τρόπο ισόρροπο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η νομοθεσία και η ανταλλαγή εμπειριών, υπάρχουν και κάποια προβλήματα ως προς τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ε, βελτιώσεις που έχουν γίνει για βάση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πλήρη εικόνα του φαινομένου ασυνόδευτων αλήκων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαβουλευτεί με τα κράτη-μέλη για να δει πώς ε, μπορούν να ε, συγκεντρώνονται καλύτερα, πιο ενιαία και πιο ε, ομοιόμορφα. Τώρα η εκτίμηση της ηλικία είναι σημαντικό θέμα γιατί είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς την ηλικία ενός ατόμου, όταν είναι ένας ανήλικος ή παιδί, ασυνόδευτος. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Η ΕΑΣΟ εργάζεται πάρα πολύ προς την κατεύθυνση αυτή και καταλήξαμε σε προτάσεις μετά από συνεδρίαση με εμπειρογνώμονες που έγιναν και διάφορα σεμινάρια. Ε, επίσης η αναζήτηση της οικογένειας είναι κάτι σημαντικό και ο εντοπισμός της για να επανέλθουν οι οικογενειακοί δεσμοί. Αυτό είναι σημαντικό για την ευημερία, για το μέλλον του ανηλίκου. Βεβαίω θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα το βέλτιστο δυνατό συμφέρον του ανηλίκου και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη βοήθεια των χωρών προέλευσης, ο εντοπισμός των οικογενειών δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκή συνεργασία με τα κράτη αυτά για την ε, πρόληψη της διακίνησης ανθρώπων και την καταπολέμηση, για την πρόληψη της ε, ε, μη ασφαλούς μετανάστευσης. Η Πρόεδρος διακόπτη. Ναι, ναι, ολοκλήρωνα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ε, δουλειά. Θα πρέπει να συνεχίσει με όλους τους ενεχομένους συμπεριλαμβανομένης της κοινωνία των πολιτών και διεθνών οργανισμών για να ε, συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα δράσης, ε, να επικεντρωθούμε στα θέματα που σας ανέφερα τα επιμέρους, τα ειδικά. Ελπίζουμε να εγκριθεί μέχρι τα τέλη του έτους το θέμα αυτό της οδηγίας του ασύλου. Συνεργαζόμαστε και με την ΑΣΟ ε, για το ερωτηματολόγιο για να ε, γίνει όσο πιο ε, καλή η αναζήτηση και ο εντοπισμός των οικογενειών. Και κατόπιν ετήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύσαμε ε, την περασμένη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μια προκήρυξη που είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου για ένα project για τους συνόδευτους ανηλίκους. Ακολουθεί η Πατή Αρμοστία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όχι για τους πρόσφυγες μάλλον λέει η Πρόεδρος. Κύριε Τζέραρτ, παρακαλώ να τηρήσετε ε, το χρόνο σας 7,5 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα αν είναι δυνατόν να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, Φιλιπ Κόλλη από τη UNICEF. Η ε, UNICEF θα μιλήσει πρώτη, αν δεν γίνεται. Μάλιστα, ακούμε λοιπόν πρώτον τον κύριο Κόρη από την UNICEF. Δεν αλλάζει όμως αυτό κάτι με το χρόνο ομιλίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε να συμμετέχουμε στις συζητήσεις σας. Ε, ήρθαμε εδώ για να σας ζητήσουμε να συνεχίσετε τις προσπαθίες σας ε, και τα όσα είπε η συγγήτρια μας βρήκε σύμφωνος και εμείς κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο ισχύει και για τη συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες γιατί εκτιμούμε ότι ένα από τους τέσσερις ετούντες ασύλου στην Ευρώπη είναι παιδιά. Αυτά είναι τα επίσημα δεδομένα που έχουμε. Φαντάζεστε ότι σε αυτό το τομέα έχουμε πολύ λίγα δεδομένα για το πώ έχει το πρόβλημα στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη. Μιλάμε περίπου για 115.000 παιδιά ετησίω. Μια τάση που παρατηρήσαμε. Η ιδέα τη σύμβαση πριν από 30 χρόνια προήλθε από το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε την ευπαθή κατάσταση των των παιδιών, τα συγκεκριμένα δικαιώματα των παιδιών. Κάποιοι είπαν γιατί να έχουμε ειδική σύμβαση για τα παιδιά αφού υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση των παιδιών και είναι σαφές ότι σε, στα πλαίσια μιας μεταναστευτικής διαδικασίας είναι ακόμη πιο τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ακόμη περισσότερο ε, τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ε, και Μπορώ να σα πω ότι αυτή η σύμβαση έχει ε, επικυρωθεί από το σύνολο των κρατών μελών, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 3 τη συνθήκη τη Λισαβόνα επίση αναφέρεται στην ε, Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Το άρθρο 3 τη ε, σύμβαση για τα Δημοκρατία των Παιδιών μιλάει για το ύψιστο σήμερα του παιδιού, όπω είπε και η συγγήτρια και το άρθρο 3 της ε, χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων επίσης. Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία για να κάνουμε κάτι. Όταν μιλάμε για το ύψιστο συμφέρον του παιδιού στο πλαίσιο της μετανάστευσης, όλες οι ερμηνείες είναι δυνατές ε, από το ένα κράτος στο άλλο και δεν μιλώ μόνο στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Μπορούμε να έχουμε και διάφορες συγκυρίες που θα μπορούσαν ε, να ισχύουν για να ε, φροντίσουμε το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Στο άρθρο 3 η σύμβαση ε, αναφέρεται στο ότι πρέπει να υπερισχύουν όλες οι δράσεις που φροντίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Στο πλαίσιο της μετανάστευσης τίθεται το πρόβλημα για το πώς τα μεταχειρίζονται αυτά τα παιδιά οι διάφορες υπηρεσίες, δημοσίες υπηρεσίες όταν ε, είναι νόμιμοι μετανάστες, όταν είναι παραμετανάστες ακόμη χειρότερα. Η ιδέα η δική μας ήταν να εργαστούμε με τους δικαστές και θα αναφερθεί ο συνάδελφος σε αυτό το θέμα, σε ένα νομικό συνέδριο με τους δικαστές ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ε, το πώς σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πώς έγινε σεβαστό το ύψιστο συμφέρον του παιδιού για να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πιο κοινέ και συνεκτικές προσεγγίσεις στο σύνολο των χωρών και να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε και εμπειρίες κατά κάποιο τρόπο. Η μελέτη, έχουμε κάποια αντίγραφα ε, που έχουν ε, διατεθεί. Πηγαίνει ακόμη πιο μακριά. Θέλουμε να δώσουμε ένα εργαλείο σε αυτό το δικαστέ σε σχέση με τη μελέτη της νομολογίας ε, Στι διάφορε υποθέσει. Δηλαδή θέλαμε να πάμε πιο πέρα από τον ότι πρέπει να υπερισχύει το ύψο στο συμφέρον του παιδιού. Προσπαθούμε να ε, έχουμε μία κοινή κατανόηση στο πόσο γίνεται σεβαστό αυτό το ύψο στο συμφέρον και να ενεργοποιήσουμε και του δικαστέ. Και αυτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο τη μετανάστευση, είτε πρόκειται για νόμιμη είτε για παράνομη μετανάστευση για μα, ένα παιδί σύμφωνα με τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, είτε είναι νόμιμο ή παράνομο μετανάστευση, έχει ακριβώ τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό θέλουμε ακριβώ να πούμε ότι ένα παιδί που και αν βρίσκεται στον κόσμο, είτε βρίσκεται σε κατάσταση μεταναστευτή, όχι ακριβώ τα ίδια δικαιώματα και δεν πρέπει να θίγονται αυτά τα δικαιώματα επειδή έχει το καθεστώς του μετανάστη ή ε, το καθεστώς ε, του μετανάστη γονιού. Ε, έτσι λοιπόν αυτό είναι σημείο που θέλουμε να προωθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και ελπίζουμε να μας βοηθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσουμε όφηση Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας είναι ένας εταίρος ε, πολύ σημαντικός και μοναδικός στο σημερινό πλαίσιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή νομοθεσία με μια ε, προσέγγιση κοινή σε όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται και για τη σεβαστό το ύψος των συμφέρον του παιδιού στο πλαίσιο της μετανάστευσης και ο συνάδελφος θα αναπτύξει περισσότερο αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σα εκ μέρου τη υπατή Αρμοστίας του ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επ' ευκαιρία της συζήτησής σας για την πολιτική για τους ασυνόδευτους ανήλικους, όπως λέτε εσείς, και όπως εμείς προτιμούμε να λέμε ασυνόδευτα παιδιά. Φυσικά δεν είναι πρόθεσή μου να επικεντρωθώ στην ορολογία, αλλά να επαναλάβω αυτό που είπε και ο συνάδελφο από τη UNICEF. Εμεί χρησιμοποιούμε τον όρο παιδιά και όχι ανήλικοι. Και αυτό διότι ακολουθούμε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που η οποία θεωρεί όλους τους ανθρώπους κάτω από 18 χρονών παιδιά, οι οποίοι έχουν, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και γι' αυτό πρέπει να προστατεύονται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τους θεωρούμε παιδιά ασχέτως από το καθεστώς νομιμότητας των ε, γονιών τους. Και οι αποφάσεις νομικές και δικαστικές που θα λαμβάνονται θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συμφώνου, να έχουν ως ύψιστο, ύψιστη προτεραιότητα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Τώρα, όπως είπε ο συναδελφό μου, ορισμένες από τις συζητήσει τη πολιτικής ανάμεσα στον εκτελεστικό και στον νομοθετικό τομέα των κυβερνήσεων παραβλέπουν τον σημαντικό ρόλο της ε, δικαστικής εξουσίας, η οποία μπορεί να ε, ανταλλάξει βέλτιστε πρακτικές και να λειτουργήσει καθοδηγητικά όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία θέτονται σε ε, κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί το καλό των παιδιών υπόψη στην νομοθετική διαδικασία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε την σοφία των καλύτερων δικαστικών ε, μυαλών στον τομέα αυτό σε όλη την Ευρώπη, από την Πορτογαλία στην Ουγγαρία και το δικαστήριο στο Στρασβούργο και να μην διατυπώσουμε γενικές συστάσεις, αλλά να επικεντρωθούμε συγκεκριμένα σε τέσσερις τομείς στους οποίους οι πρακτικές είναι διαφορετικές και προβληματικές. Αυτή η τομείς ήταν η ηλικία, οι διαδικασίες αξιολόγησης, οι βιώσιμες λύσεις, για παράδειγμα, οι αποφάσεις, η πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές παροχές και άλλα κοινωνικά δικαιώματα και δικονομικές ε, ασφαλιστικές τυκλίδες και υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις, ε, στη νομική παράδοση των κρατών μελών αλλά και στις ε, πρακτικές. Υπήρχε ένας μεγάλος βαθμός συνένεσης ανάμεσα στους δικαστές σχετικά με το πώς θα εφαρμόζονται οι αποφάσεις για το καλύτερο συμφέρον των παιδιών και οι δικαστές βρήκαν πώς μπορούν να εφαρμοστεί αυτό οι βέλτιστε δηλαδή πρακτικές ε, ε, στην ισχύουσα κατάσταση στα κράτη-μέλη. Και αυτές οι καλές πρακτικές υπάρχουν τώρα, αλλά υπάρχει ασυνέπεια στα κρατη ε, όχι ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη, στο ίδιο το κράτος μέλος. Να σας δώσω μία σύντομη τώρα περίληψη. Όσον αφορά την αξιολόγηση της ηλικίας, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη, είτε ιατρικές, είτε κοινωνικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις και η μία αποκλείει την άλλη και δυστυχώς αυτή που υπερισχύει είναι η πιο αρνητική αξιολόγηση και αυτό εξαρτάται από την νομική παράδοση και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Ε, συμπεράναμε λοιπόν ότι όλες οι μέθοδοι ε, ε, υπολογισμού της ηλικία έχουν, έχουν μεγάλα περιθώρια λάθους, καμία από αυτές όμως δεν επαρκεί. Και όταν έχουμε στοιχεία από εμπειρογνώμονε τα οποία δεν συμφωνούν, τότε πρέπει ο ανήλικό να θεωρείται παιδί. Η απόφαση να είναι προ όφελό του και πρέπει να υπάρχει επίση η ευκαιρία να γίνεται ένσταση ενάντια τη εκτίμηση της ε, ε, ε, εκτίμησης και να υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στην δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις βιώσιμες λύσεις τώρα, οι καλές, πρακτικές, οι καλές δικαστικές πρακτικές για τους ασυνόδευτους ανήλικους συμπεριλάμβαναν διοικητικές αποφάσεις επιστροφής των ανήλικων χωρίς και δαιμόνα στη χώρα προέλευσης. σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ε, άλλα μέλη της οικογένειας ή άλλοι διακανονισμοί, το δικαστήριο ζήτησε να επιστρέφεται, όταν επιστρέφεται το παιδί στη χώρα προέλευσης, να υπάρχει μια ξεκάθαρη αιτιολόγηση και ταυτόχρονα να λαμβάνονται υπόψη τα βελτιστά συμφέροντα του παιδιού. Προτάθηκε λοιπόν να επιστρέφεται το παιδί στη χώρα προέλευσης εάν και μόνο εάν διασφαλίζεται το καλό του παιδιού και εντοπίζεται η οικογένεια. Διαφορετικά το παιδί και, και επίσης το παιδί σε καμία περίπτωση να μην επιστρέφεται σε χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Επίσης, έπρεπε να ζητήσουμε ε, ότι οι αρμόδιες αρχές ε, πρέπει να παρέχουν κυδαιμονία στο παιδί και να του επιτρέπουν να αποκτήσει άδεια παραμονής και να μην έχει το καθεστώς παράνομου μετανάστη. Έχουμε το, το... Ε, έχουμε παιδιά τα οποία μέχρι τα 18 του χρόνια βρίσκονται σε καθεστώ προστασία και με το που κλείσουμε το που ενηλικιωθούν θεωρείται παράνομοι μετανάστε. Και αυτό φυσικά Και όσον αφορά το κέντρο κράτηση, θεωρήθηκε ότι δεν είναι στο, στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να, υπάρχει, να οδηγείται σε κέντρο κράτηση ε, μαζί με ενήλικες. στη συμφωνία με το άρθρο 31 του συμφώνου και επίσης όταν, τα, όταν οι συνόδευτοι ανήλικοι φτάσουν τα 18 έτη να έχουν τις, τα ίδια δικαιώματα για ιατρική περίθαλψη. Έπειτα, ασφαλιστικέ δικλείδε. Το δικαστήριο εντόπισε βέλτιστε πρακτικέ, οι οποίε συμπεριλαμβάνουν το ότι ένα παιδί πρέπει να ε, έχει κάποιον ε, κηδεμόνα διορισμένο από τη στιγμή που ε, αναγνωριστεί ως ασυνόδευτο ότι το παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τη δική εκδοχή των γεγονότων και να έχει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή του στο δικαστήριο, γιατί αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του. Και επίσης το παιδί έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση και η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης να γίνεται με βοήθεια. Επίσης, οι αρχές που ασχολούνται με μεταναστευτικά ζητήματα πολύ συχνά παραμελούν τα συμφέροντα των παιδιών. Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής ε, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και πραγματικά θα χαιρόμασταν πολύ εάν βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθεί η δική μας έκθεση στην πρότασή σας. Είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και μπορείτε να τη διαβάσετε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουν γραφεί 5, 6, 7 συνάδελφοι, 8 τώρα για τη συζήτηση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ πρώτη. Ευχαριστώ Σοφία. Καταρχά θα ήθελα να πω ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομη διότι η συγγήτρια Αναταλή ε, Γκρισμπέκ και οι συνάδελφοι τη UNICEF και του ΟΗΕ τη ΥΠΑ τη Αρμοστία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέδειξαν ποιε είναι οι προκλήσει τα προβλήματα και οι περιπλοκές ε, σε θέματα ανηλίκων παιδιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σκιώδη συγγήτρια από πλευρά του ΕΛΚ γιατί πρόκειται για 75.000 παιδιά, 75.000 παιδιά που φτάνουν χωρίς τους γονείς τους σε ένα νέο κόσμο και είτε είναι θύματα πολέμου, σύραξης ή ακόμα και ε, διακινητών που τους έχουν ε, πουλήσει αγοράς. Είναι πρόβλημα ανθρώπινο και ψυχολογικό. Έχουμε μια πολύ καλή βάση πάντα στις εκθέσεις μας να συζητάμε ε, με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα του, του Κοινοβουλίου συγγνώμη, στο πακέτο του ασύλου και χαίρομαι που πέρασαν οι τροπολογίες μας ε, στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης ε, και που αναγνωρίσαμε ακριβώς το ύψιστο ε, συμφέρον του παιδιού ως τμήμα της δική μας νομοθεσίας. Το θέμα της νομικής εκπροσώπησης, ε, ερμηνείας ειδική εκπροσώπησης και στην οδηγία για τις κακοποιήσεις των παιδιών, όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι χαίρομαι πολύ και καλωσορίζω το γεγονός ότι είναι πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη και προσανατολισμένη σε δράση η πρόταση της εισηγήτριας. Είναι πολύ συνεκτική η έκθεση και μπορούμε να βελτιώσουμε και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Βασικά εμεί έχουμε τώρα στοιχεία μόνο για τους ετούντες άσυλο και δεν υπάρχει μία λύση ε, ενιαία που να εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά που φτάνουν στην Ευρώπη. Χρειάζονται μέτρα ad hoc, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερο ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, γιατί έρχονται, ποια είναι τα κίνητρά τους. Και αν δεν ζητούν άσυλο, τι θα γίνει. Στη Σουηδία, μόλις ε, μόνο το 2011 ήρθαν 2.655 παιδιά και είναι ο πιο ε, ψηλό αριθμό στην Ευρώπη με τάση αυξητική. Γι' αυτό ε, υπάρχει πρόταση να έρθει η Επιτροπή μα να κάνει μια επίσκεψη και ελπίζω να το εγκρίνουν οι συντονιστές ότι ακόμα και σε μια χώρα που λειτουργεί το σύστημα είναι τεράστια τα προβλήματα και οι προκλήσεις. Γιατί σε τελική ανάλυση οι δήμοι και οι κοινότητε. Ε, είναι ο σωστός τόπος να εξεταστεί αυτό. Οι οικογένειες, η συνένωση των οικογενειών είναι το σωστό μέσον. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρακτικά ζητήματα που πρέπει να μελετήσουμε και ελπίζω να έρθετε στη Σουηδία να ανταλλάξουμε ε, βέλτιστες πρακτικές και να δείτε και τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας ε, κακοποιώ, αλλά πρέπει να σας πω ότι καθένας έχετε δύο λεπτά για να μιλήσετε, αλλιώς δεν θα προκάνουμε. Συγγνώμη, λέει η κυρία Κοράτσα, εκτό μικροφώνου, αλλά πρέπει να τα πω. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχουμε σκιώδει ηγητέ, αλλά και οι σκιώδει ηγητέ ομιλητέ είναι. Και μία ώρα είναι 60 λεπτά μέχρι νεοτέρα. Οπότε είτε είστε σκιώδει είτε δεν είστε, πρέπει να χωρέσετε. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ακούσαμε πάρα πολύ ότι στο κέντρο θα πρέπει να είναι το παιδί και τα συμφέροντα του παιδιού, να είναι το υπαριθμό να ένα ζητούμενο πριν από οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Βλέπω όμως την κατάσταση στα κράτη-μέλη και απέχει πόρο από την πραγματικότητα να είναι ε, στο επίκεντρο η ευημερία του παιδιού. Ακόμα και ασυνόδευτοι ανήλικοι παιδιά μεταναστών θεωρούνται πρόβλημα, πρόκληση, ε, παράγον κόστους. Και καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι ε, έχει σημασία ε, η εκτίμηση της ηλικία, ο υπολογισμός για να δούμε αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα κρατήσουμε ή αν επιτρέπεται να τα στείλουμε πίσω. Ακούστηκε επανειλημμένα το πακέτο του ασύλου, αλλά θέλω να ξαναπώ ότι αν πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει και αυτός ο συμβιβασμός που έχει βρεθεί μέχρι τώρα γιατί δεν έχει καταλήξει να είναι διαφορετικός από αυτό που ισχύει τη στιγμή και τα επόμενα βήματα που έχουν σκεφτεί δεν νομίζω ότι έχουν ως γνώμονα το συμφέρον του παιδιού σε πρώτη βάση, αλλά θέλουν να αποφύγουν να έρθουν παιδιά. Και αν έρθουν το συντομότερο να μπορέσουμε να τα στείλουμε πίσω. Θα πρέπει να ενημερώνονται, λέτε, στις χώρες προέλευσης για το πόσο επικίνδυνη είναι η μετανάστευση. Γιατί, για να μην φεύγουν τα παιδιά. Μα τα παιδιά που φεύγουν ξέρουν πολύ καλά τι κινδύνους διατρέχουν. Και ποια οικογένεια στέλνει τα παιδιά της έτσι. Και η συνένωση των οικογενειών βεβαίως είναι κάτι ε, που μας απασχολεί και ακούσαμε ότι τουλάχιστον σε περιπτώσεις εμπόλεμων χωρών να μην στέλνουμε παιδιά πίσω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι καταστάσεις, θεομηνίες, λοιμοί, όπου δεν υπάρχει ε, δυνατότητα ή δεν είναι ιδεώδης κατάσταση να συνενωθεί η οικογένεια σε ένα τέτοιο τόπο. Και θα παρακαλούσα τελευταία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μου πούν τι εστί πρόληψη ανασφαλούς μετανάστευσης, αν η κατάσταση στις χώρες τους είναι τέτοια ώστε δεν έχουν άλλη ευκαιρία ή δεν βλέπουν άλλη τύχη και ποιες είναι πραγματικά οι φόρες λύσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες προέλευσης ε, για τα παιδιά των μεταναστών. Και τελικά η μετανάστευση να μην χρειάζεται που είναι και πάντα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκεί νομίζω κάνουμε πολύ λιγότερα ε, από τα άλλα για τον προσδιορισμό της ηλικία για την ενημέρωση για τον κίνδυνο. Η σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε το χρόνο σας, γιατί θα χτωθούμε εδώ πέρα, κυρία Φλότρο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι... Πώς να το πω... Είναι λίγο απογοητευτικό. Πρώτη συζήτηση για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα και οι σκιώδεις συζήτητες, ενώ είναι πάρα πολύ ε, ε, ισχνή η ε, παρουσία των βουλευτών και οι σκιώδεις να μην έχουν δύο λεπτά. Ορίστε, έχασα 15 δεύτερα και έχω ένα και 45 τώρα. Εγώ ε, βλέπω ότι είναι πολύ θετική η βάση για τη συζήτηση αυτή και η Ιωνή. Η κυρία Κρισπέκ πραγματικά το έχει θέσει στα σωστά θεμέλια, έχει τονίσει όλα τα σημαντικά ερωτήματα στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε και το θέμα πολύ εύστοχο ε, του νέου καινοτόμου και στοχευμένου νομοθετικού μέσου για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ή ε, έλλειψη συνέπειας ε, και το ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την UNICEF και από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολύ εύστοχο τρόπο. Για τα αριθμητικά στοιχεία, από ό,τι φαίνεται η πολιτική μας ε, και ε, τα νομοθετικά μέσα που έχουμε για την προστασία των παιδιών έχουν ε, πάρα πολλά παραθυράκια. θέλετε είναι ένα δίχτυ που έχει πάρα πολύ μεγάλα μάτια και περνάνε από εκεί και χάνονται και ανηλικοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μιλάει για 16.631 ασυνόδευτους που ζητούν άσυλο και έχουν λάβει άσυλο για την Ευρώπη των 27 οι ενώσεις και τα σωματεία μας λέγουν ότι στη Γαλλία μόνο είναι 8.000 ε, μεμονωμένοι και ασυνόδευτοι ανήλικοι και προσπαθούν να ε, νομιμοποιηθούν είτε με το άσυλο είτε άλλος πώς, αλλά εκκρεμούν ακόμα αυτές οι υποθέσεις. Ε, στη συνέχεια, ε, ποια είναι τα νομοθετικά μέσα που έχουμε. Θα πρέπει να τα καταστήσουμε πιο συνεκτικά στο πακέτο για το άσυλο, τα θέματα της δικονομίας και της διαδικασίας. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα με το Συμβούλιο να αποφύγουμε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να εξαιρούνται από όλες τις ε, εξαιρέσει και τις παρακάμψεις των διαδικασιών και ακόμα και η ίδια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ περιοριστική σε αυτό το τρίπτυχο πρόληψη, υποδοχή, βιώσιμη λύση. Ακούμε ότι η βιώσιμη λύση είναι καταρχήν επαναπροώθηση. Εγώ ε, θέλω να σας παραπέψω στον εκπρόσωπο του ΟΗΕ για αυτό το ζήτημα. Ξέρω ότι τέλειωσε ο χρόνος μου. Χαίρομαι για την έκθεση. Είμαι στη διάθεση της ηγήτριας και θα βάλω όλοι μου τα δυνατά για να εγκρίνει το πιο καλό και το πιο χρήσιμο κείμενο του Κοινοβούλιο για την προστασία των ανηλίκων. Ευχαριστώ κυρία Φλότρου και εγώ αισθάνομαι την ίδια ματέωση και απογοήτευση. Μπορεί κανείς να μας προτείνει πώς μπορούμε να βάλουμε 120 λεπτά σε μία ώρα, τότε θα μιλήσετε περισσότερο. Ο κύριος Μπρόνς, επόμενο στον κατάλογο μου. Ε, ευχαριστώ. Άρθρο 3 το ύψος του συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Αυτά έχουν γραφτεί σε μάρμαρο. Μπορούν να αλλάξουν. Θνητοί τα έχουν δώσει και όχι ο Θεός και μπορούν να τα αλλάξουν οι θνητοί. Τα, οι ανήλικοι έρχονται συνόδευτοι στην Ευρώπη για ποιο λόγο. Υποθέτω ότι είναι αντικείμενο διακινητών δολίων και ορισμένοι όμως έχουν παραπλανηθεί ε, από κάποιους που καλή την πίστη τους παραπλάνησαν. Ποιο είναι το υλικό συμφέρον του παιδιού. Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί. Ε, μάλλον, ε, ε, μπορεί το παιδί να ζει καλύτερα στην Ευρώπη οικονομικά από πλευρά ευημερία, αλλά αποκόπτεται από τις ρίζες του. Και είναι πολύ σημαντικό ε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πέρα από την προέλευση και το ε, πολιτιστικό του υπόβαθρο, τι κάνουμε με τα παιδιά. Ε, αναρωτιόμαστε αν μπορούν να παραμείνουν στον τρίτο κόσμο ασυνόδευτα ή συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους. Μήπως να τα φέρουμε όλα στην Ευρώπη. Και είπαμε να, να εξηγούμε και στους συνοριοφύλακες πώς θα του φέρονται και πώ θα τους υποδέχονται. Μήπως να τα πούμε στα μέλη της Επιτροπής μας όλα αυτά για να συνετιστούν. Τουλάχιστον ε, τήρησα το χρόνο μου, αν μη τι άλλο, η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι εμεί αυτήν την αίθουσα, νομικοί που ασχολούμαστε με θέματα σχετικά με παιδιά, συμφωνούμε πλήρω ε, με την αρχή ότι το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να ε, βρίσκεται σε πρώτη θέση, είτε μιλάμε για υπόθεση της ύφεσης της κάγης είτε μιλάμε για μια υπόθεση συνοδευτού ανηλικού μετανάστη, αλλά το ζήτημα είναι ποιο ακριβώς είναι το συμφέρον του παιδιού και ποιος το αποφασίζει αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Κορατσαμπίλ το ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά ερωτήματα αν θα πρέπει να επαναπατρίζεται ένα παιδί ή όχι, αλλά δεν συμφωνώ ότι αυτά είναι πρακτικά ερωτήματα. Αυτά δεν είναι πρακτικά ζητήματα, είναι θεμελιώδη ζητήματα αρχής και θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές για τη δικαστική πρακτική, για το αν ε, υπάρχει τεκμήριο ότι ένα παιδί από τον τρίτο κόσμο πάντοτε είναι προς το βέλτιστο συμφέρει του να παραμείνει στο δυτικό κόσμο και ναι, γιατί. Και ποια είναι η αρχή και ποιο είναι το σύστημα αξιών και η αιτιολογία πίσω από αυτό. Επίσης, μας είπαν ότι σε μία υπόθεση παραβίασης ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε μία φυσικά σωστή απόφαση από το δικαστήριο γιατί υπήρξε κράτηση ενός παιδιού πέντε μηνών και ενός παιδιού τριών ετών σε ένα κέντρο κράτησης. Αλλά Ουσιαστικά, ποιε είναι οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από δεκάδες χιλιάδες ιστορίες της ΙΟΣ και ποια είναι η ακριβώς Ποια είναι ακριβώ η νομική διαδικασία, ποιο εκπροσωπεί αυτά τα παιδιά, ποιε ε, είναι οι αρχέ και ουσιαστικά πώς ε, κρίνεται το βαλιστό συμφέρον του παιδιού όταν ε, λαμβάνεται η απόφαση αν ε, θα επιστραφεί το παιδί ή όχι. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτά τα θέματα, κυρίως γιατί στην τεκμηρίωσή μας δεν βλέπω, δεν ε, βλέπω να γίνεται αναφορά σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Μπάρ. Ευχαριστώ. Έχω να προσθέσω δύο ερωτήσεις. Σίγουρα η εκτίμηση της ηλικία είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο, όπως υπόθηκε. Σε πολλές περιπτώσεις ε, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η ηλικία των παιδιών ε, είναι και εξευτελιστική. Αυτές οι μέθοδοι είναι πάρα πολύ παλιές. Μιλάμε για μεθόδους ε, που ε, μπορεί να χρονολογούνται 100 έτη πριν. Ε, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να συμμεθεί κάποια πρόοδο σε αυτό το θέμα. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την εμπορία ανθρώπων. Είναι μάλλον μια ερώτηση που σχετίζεται και με την εμπορία ανθρώπων. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά σήμερα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι έμποροι του, τα φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έμποροι ε, ανθρώπων όμως ε, δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε. Υπάρχουν και παιδιά που έρχονται μόνα τους και βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υπάρχουν πάρα πολλά θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 1 τέταρτο των θυμάτων είναι παιδιά. Έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερα περίεργη κατάσταση. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδιών που έρχονται από τρίτε χώρε, αλλά δεν ανησυχούμε με τον ίδιο τρόπο για τα παιδιά που ε, φτάνουν σε όλα κρατημέλη από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω πώ θα λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποια σχετική ιδέα. Ευχαριστώ κύριε Μακεντέρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι κάθε συνόδευση συνολικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρείται παιδί και να υπάρχει και ανάλογη μεταχείριση και ότι πρέπει να έχουμε κατά νου το περισσότερο συμφέρον του παιδιού. Επίση, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τα καλύτερα δυνατά πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τι πληροφορίε που μα έδωσε σήμερα. Αυτό που με εκπλήσει είναι το εξή. Νομίζω ότι σε ορισμένε ε, χώρε δεν γίνονται σεβαστέ υποχρεώσει ε, που έχουν αναλάβει δυνάμει τι συνθήκε. Ε, και εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχέδιο, απλώ δράση χρειάζεται. Και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι κάνει αυτή για να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη σέβονται τι υποχρεώσει του δυνάμει των συνθήκων. Η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω αφορά το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Το σχέδιο δράσης να τα κράτη-μέλη να ε, καταρτήσουν ε, τους ε, αρμόδιους και να βοηθήσουν τους συνεροφυλακές να κάνουν τη σωστή εκτίμηση. Έτσι λοιπόν, μήπω η Κομισιόν θα μπορούσε να μα δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία για αυτή την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση και πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τι διαφορές μεταξύ ενό παιδιού που είναι υπεμπειρία και ένα παιδί που ε, είναι χωρίς επίτροπο και ζητά άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι οι εκατοντάδες παιδιά είναι αντικείμενο εμπορία ετησίω και τα μισά από αυτά καταλήγουν και πάλι πίσω στου ανθρώπου που τα έχουν εχμαλωτήσει. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε ότι ακόμη και αν τίθενται υποφροντίδα, αυτά τα παιδιά φοβούνται τόσο πολύ και τελικά καταλήγουν με του ανθρώπου που αρχικά τα εκμεταλλεύονται. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ και ο κύριος Τρεντεφιλίδη είναι ο τελευταίος ομιλητής. Και εγώ, Πρόεδρε, είμαι πολύ ευγνωμών στην εισηγήτρια και τους υπολείπους που υπογράμμισαν τα βασικά ζητήματα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς αυτό το θέμα. Τα σερούμε αυτά τα παιδιά μετανάστες ή παιδιά γιατί για παιδιά δεν τίθεται θέμα κέντρων κράτησης, ούτε επαναπροώθησης, ε, ούτε μετεγκατάστασης. Εάν τους βλέπουμε ως μετανάστες, τότε έχουμε όλες αυτές τις έννοιες στο μυαλό μας, που συνδέονται με μετανάστες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω θέματα που ήδη αναφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσβαση υπηρεσίες πρόσβαση ε, ακριβώς νομική φροντίδα και στέγη, τροφή, εκπαίδευση, μόρφωση. Μέχρι τώρα δεν ακούστηκαν. Προσβλέπω λοιπόν ε, στην έκθεση της εισηγήτριας για να δούμε πώς αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και πώς θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και εγώ, ιδιαίτερα για το ότι ήσασταν σύντομος. Κάποιες απαντήσεις Κάποιε ερωτήσει μάλλον απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αντιπρόσωπους του ΟΗΕ και τη UNICEF. Θα ήθελα να ρωτήσω από τον καθένα από αυτούς να τους ζητήσω να απαντήσουν πολύ σύντομα. Το πολύ δύο λεπτά ο καθένας, εκτός αν δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα, κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντως, πολλές οι ερωτήσεις που έγιναν και αυτό τι καταδεικνύει ότι Όλες οι ερωτήσεις αυτές που συνδέονται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους δεν είναι εύκολες στην επίλυσή τους. Ρώτησε και η κυρία Σίπελ τι κάνουμε ακριβώς στις χώρες ε, ε, καταγωγής τους. Βεβαίως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ανήλικοι έρχονται για διάφορους λόγους. Ορισμένοι θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, άλλοι αντιμετωπίζουν δύσκολη κατάσταση και ζητούν άσυλο και είναι άλλη κατάσταση αυτή από τους ανηλίκους που φτάνουν εδώ για λόγους οικονομικούς ή για λόγους που συνδέονται με την ένδυα, με την έλλειψη παιδείας και έρχονται να βρουν καλύτερο κόσμο στην Ευρώπη. Επίσης, όχι οι ανήλικοι που έρχονται για λόγους πολέμου, αλλά για τους άλλους θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε στα πλαίσια της ε, ε, αναπτυξιακής συνεργασίας στις ε, πατρίδες τους για να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Η κατάσταση των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίου ανθρώπων είναι και αυτή γνωστή και έγιναν πολλές ερωτήσεις σχετικά θα ήθελα και πάλι να σας παραπέψω στην πρόσφατη οδηγία που εγκρίθηκε για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που ε, αναφέρεται ρητά στο ύψος του παιδιού και περιλαμβάνει και διατάξεις που ελπίζουμε να μεταφερθούν σε εθνικές νομοθεσίες από τα κράτη-μέλη και μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει το ρόλο της θεματοφύλακα των συνθηκών και θα παρακολουθεί την εφαρμογή των οδηγιών. Όχι μόνο για τούτη εδώ την οδηγία, αλλά και για την άλλη και οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται με την οδηγία αυτή είναι ήδη σε επαφή με τα κράτη-μέλη για να γίνει όσο γίνεται καλύτερα μεταφορά, αλλά και για τι άλλε οδηγίε που ήδη ισχύουν για το άσυλο, α πούμε, και εκείνες που πρόκειται να εγκριθούν και ε, να μεταφερθούν ε, σύντομα στι εθνικέ νομοθεσίε. Για να απαντήσω σε μία λοιπόν από τι ερωτήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει το ρόλο τη θεματοφύλακα των συνθήκων και θα κινήσει διαδικασίε επί παραβάση αν χρειάζεται ε, αν ε, θεωρεί ότι υπάρχει από χρόνο λόγος. Κάτι που αναφέρθηκε για τις βιώσιμες λύσεις. Δεν νομίζω ότι βιώσιμη λύση αυτή καθ' αυτή είναι η επαναπροώθηση. Θα πρέπει να γίνει σαφέστατα πάντα η διάκριση. Για ποιο λόγο έρχονται εδώ, αν είναι τον άσυλο, ε, δεν είναι λύση η επαναπροώθηση, θα πρέπει να τους δίδεται διεθνής προστασία. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε, λέει η Πρόεδρος. μάλιστα. Επίσης αναφερθήκαμε στο πρόγραμμα δράσης μας ε, στη πιθανή ε, ένταξη των παιδιών αυτών εδώ στην Ευρώπη. Και αποφασίσαμε να τα υποστηρίξουμε μέσω του Ταμείου της Ένταξης. Δυστυχώς κανένα κράτος μέλος δεν έκανε χρήση αυτού του χρηματοδοτικού μέσου μέχρι σήμερα. Και από την άλλη δεν θα πρέπει να αποκλείεται πλήρως η επιστροφή, γιατί κανονικά ένα παιδί αισθάνεται καλύτερα στην οικογένειά του. Ε, Αυτά είναι μερικά στοιχεία. Είμαι στη διάθεσή σας και για διμερείς απαντήσεις. Είμαι βεβαίω ότι θα έχουμε και άλλη ευκαιρία για συζήτηση, αλλά έχουμε και άλλη συζήτηση που ακολουθεί, γι' αυτό θα σας περιορίζω. Ο κύριος Κόρη και μετά ο κύριος Τζεραπ. Δύο λεπτά το πολύ έκαστος. Θα μιλήσω εκ μέρους και των δύο μας, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά την επιστροφή διατυπώθηκε το ερώτημα εάν κάτω από το καλύτερο συμφέρον του παιδιού εννοούμε ε, το ότι δεν πρέπει να επιστρέφεται κανένα παιδί. Όχι, δεν εννοούσαμε αυτό. Δεν συμπέρανε αυτό το δικαστικό συνέδριο κάτω από τις ε, βέλτιστες πρακτικές και τις βιώσιμες λύσεις. Θεωρείται ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι να επιστρέψει και να ζήσει με τους γονείς του στη χώρα προέλευσης όπου οι γονείς θα μπορούν να του προσφέρουν την κατάλληλη βοήθεια. Αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου οι αρχές προσπάθησαν να επιστρέψουν παιδιά σε περιπτώσεις οι οποίες απορρίφθηκαν μετά από τους ε, δικαστές. Για παράδειγμα, περιπτώσεις όπου δεν είχαν γίνει διακανονισμοί για την υποδοχή, όπου δεν είχε εντοπιστεί η οικογένεια και όπου δεν ήταν σαφές ποιος αξιολόγησε ή ποιος παρέλαβε το παιδί και πολλέ φορέ περιπτώσει όπου τα παιδιά επέστρεψαν σε χώρε που βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αυτέ οι περιπτώσει είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τι ε, δούμε και δεν μπορούμε να... Ε, ε, να πούμε ότι είτε δεν θέλουμε να επιστρέψουμε κανέναν, είτε να επιστρέφουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται. Όχι, πρέπει να αξιολογούμε την κάθε περίπτωση με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και με μονομένα. Όχι με φορμαλιστικό τρόπο, αλλά ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος, κύριε Κορή. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Απλώς να σας πω ότι κάναμε κάποιες μελέτες στη Γερμανία σε σχέση με παιδιά που είχαν επαναπατριστεί στο Κωσυβοπέδιο για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν πρόκειτο για την ορθή απόφαση. Εξετάσαμε πώ ήταν η κατάσταση των παιδιών αυτών πριν από την αχώρησή του στην Γερμανία. Πήγαιναν σχολείο και ήταν υπό προστασία και βρέθηκαν στο Κωσυφοπέδιο, μια χώρα που δεν γνώριζαν καθόλου, δεν μιλούσαν τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν βρίσκονταν σε μια πολύ μεγάλη κατάσταση επισφάλεια. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε δεδομένα για τέτοιε καταστάσει. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκρίσπεκ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σοφή. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αλλά και για την πολύ συγκεκριμένη απάντηση που δόθηκε στις ερωτήσεις των συναδέλφων και ευχαριστώ και ε, τους ομιλητές από το Γραφείο της Επατσιμασίας των ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και όλους τους συναδέλφους για τις προστάσεις τους τις ουσιαστικές στους μήνες που θα ακολουθήσουν ε, θα εργαστούμε σκληρά γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα και μας αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Εκτιμώ ιδιαίτερο αυτή την ιδέα που μας προτείνεται να μιλάμε συστηματικά για παιδιά και όχι για ανηλίκους. Ε, είναι ε, φορτωμένος με συμβολισμό όρος γιατί νομίζω ότι είναι προβληματικός όρος του ανηλίκου και ό,τι και να γίνει το παιδί είτε είναι σε κατάσταση παράνομης νόμισης μετανάστευση. πρέπει να θεωρούμε ότι καταρχήν είναι παιδί και έχουμε καθήκοντα απέναντι του. Για οποιοδήποτε λόγο λοιπόν ε, ήρθε ε, το παιδί αυτό αποτελεί, ε, εν να σας πω, ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τους λόγους για τους έφυγε το παιδί. Μπορεί να υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, διάφορες τραυματικές εμπειρίες. Και αυτοί που πιστεύουν ότι ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ελντοράντο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το πιστεύουν, ε, ή γιατί τι μπορείτε τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στην Ευρώπη για την αντικείμενο εκμετάλλευση, αντικείμενο εμπορία. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα θέματα πρέπει να απαντήσει η δική μας έκθεση και μου άρεσαν και όσο υπογράμμισε η Άννα Μαρία ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές δυσκολίες και ερωτηματικά που τίθενται. Και επίσης και αυτό που υπενθύμησαν οι συνάδελφοι ότι η κατάσταση είναι επίγουσα. Και υπάρχουν οι τις πρακτικέ, ίσως ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή των δεδομένων, έχουμε και ένα πιλωτικό σχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή, αλλά πρέπει να δώσουμε και συγκεκριμένε απαντήσει. Και ίσως θα πρέπει να οδηγήσουμε και τα κράτη-μέλη στο να σέβονται τις υποχρεώσει του. Και θέλω να ολοκληρώσω, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου θα έπρεπε να ε, λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία της νομολογίας. Ελπίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα συνεκτικό, κάτι που ζητήθηκε από όλους τους συναδέλφους. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Συγήτρια και περνάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Έχουμε λιγότερο από μία ώρα για τη συζήτηση για το δέσμη μέτων προστασίας των δεδομένων. Είναι ένα σημαντικό θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους εκτός της αιθούσης, παρακαλώ. Έχουμε δύο εισηγητές. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας και την νομική υπηρεσία. Και κατόπιν θα έχουμε και συζήτηση. Επομένως θα επιμείνω στην αυτοπιθαρχία. Σας παρακαλώ, αν ε, δεν δείξετε αυτοσυγκράτηση στον χρόνο, θα είμαι ακόμη πιο σκληρή. Και ήδη ανακοινώνω ότι για τη συζήτηση μόνο δύο λεπτά χρόνο ομιλίας το πολύ θα έχετε. Δύο λεπτά, όχι δύο λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Και θα ζητήσω και από τους συζητητές και από την Κομισιόν και από την Κυπριακή Προεδρία και από την Νομική Υπηρεσία να είναι πάρα πολύ σύντομοι να ξεκινήσω με τους δύο συγητές. Ε, καταρχήν ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ, Σόφη. Ε, νομίζω πως μπορώ να μιλήσω λίγο παραπάνω από δύο λεπτά. Να μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Όποιος θέλει να κουβεντιάσει, παρακαλώ να καταλήψει την αίσθουσα, έτσι ώστε να συγκεντρωθούμε στο πακέτο προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιστρέφω στον επόμενο κύκλο ανταλλαγής απόψεων για το πακέτο προστασίας δεδομένων, τον κανονισμό και την οδηγία. Ακόμα δουλεύουμε πολύ σκληρά με τους σκιώδες εισηγητές για τον φάκελο αυτό και ο κύριος Δρούτσας, ο εισηγητής της οδηγίας και εγώ αναμένουμε ακόμα να αποφασίσουμε την προσέγγισή μας για μία για ένα συνεπές καθεστώς προστασίας δεδομένων. Όπως γνωρίζετε αυτό φυσικά είναι μια μεγάλη πρόκληση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε και να το καταφέρουμε μάλιστα σε ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί να ανταπεξέλθει στο στόχο μας, να τελειώσουμε δηλαδή πριν το τέλος του χρόνου όσον αφορά τον κανονισμό. σας, έχει, σας έχουν μοιραστεί τα δύο έγγραφα εργασίας για τον κανονισμό, το υπαριθμόν 2 και το υπαριθμόν 3. Θα ήθελα να σκιαγραφήσω τα βασικά σημεία στα έγγραφα αυτά, διότι από αυτά φαίνεται πού βρισκόμαστε στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ για τον κανονισμό. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε όλο τον φάκελο, να δούμε όλες τις απόψεις και έχουμε διατυπώσει ήδη κάποιες ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε. Επίσης, όσον αφορά την έκθεσή μου, θα ήθελα να την παρουσιάσω πριν τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε όλοι να έχουν χρόνο μετά τα Χριστούγεννα και στα αρχές του 2013, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, να τη διαβάσουν καλά, να δουν όλες τις τροπολογίες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στην Επιτροπή Λύπη περίπου στο τέλος Απριλίου για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Όσον αφορά την ουσία τώρα, ένα από τα σημαντικότερα σημεία που επιθυμούμε να επιτύχουμε και θα το τονίζουμε αυτό συνέχεια. Θέλουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων του ατόμου, ενίσχυση της ε, διάστασης της εσωτερικής αγοράς και των κανόνων για την προστασία δεδομένων και ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης. Το των λεχθέντων είναι από τα κύρια σημεία όπου θα θέλαμε να δούμε εξελίξεις, είναι η ενδυνάμωση των κύριων αρχών μας. Θα θέλαμε λοιπόν ο κανονισμός να έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογή όπως η οδηγία. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η ορισμή των δεδομένων και της προστασίας δεδομένων. Θα θέλαμε λοιπόν να εναρμονίσουμε περαιτέρω τις αρχές αυτές με εκείνες που είχαμε πριν, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε το σημείο που βρίσκεται ο διαχωρισμός και τα δεδομένα, τα οποία δεν καλύπτονται από αυτό το σχέδιο προστασίας, αλλά επίσης και να τονίσουμε ότι υπάρχει κίνητρο στον κανονισμό αυτό για περαιτέρω συγκεντρωτικούς όρους και να δοθεί η ευκαιρία οι διαδικασίες να μπορούν να γίνουν περισσότερο ανώνυμες. Είτε με ψευδόνυμο. Έπειτα, το άλλο σημαντικό είναι το ζήτημα της νομικής βάσης που έχουμε για τη διαδικασία. Υπάρχει επιθυμία να υπάρχει συνένεση και για την επεξεργασία δεδομένων, αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του κανονισμού αυτού. Θέλουμε να υπάρχει προβλεψιμότητα για τα δεδομένα. Θέλουμε την ανάμιξη αλλά και την συνένεση για παροχή πληροφοριών και οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να είναι εκτενείς αλλά να είναι εύκολα κατανοητές, να μην είναι πάρα πολύ τεχνικές έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η επεξεργασία τους όσον αφορά το νομικό υπόβαθρο. Και τα νόμιμα συμφέροντα. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αύριο θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνεδρίαση άλλης επιτροπής για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να έχουμε απαντήσεις τώρα αντί να το αφήσουμε αυτό για καταξουσιοδότηση πράξης. Κάτι άλλο που θα ήθελα να θίξω, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ καιρό τώρα, αλλά να σας επιστήσω την προσοχή στα ζητήματα privacy by design, και τα ζητήματα πιστοποίησης, privacy by certification, πρέπει να προβλέπονται δυνατότητες διευκρίνησης από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Και ίσως να υπάρξει κάποια προκήρυξη για καλύτερη πιστοποίηση στην Ευρώπη. χρειάζεται να βρεθούν καλύτερες λύσεις όσον αφορά την ε, προστασία δεδομένων, ιδιαίτερα στον τομέα της πιστοποίησης. Και εδώ έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Τώρα δεν μπορώ να σας ε, αναφέρω όλες τις πτυχές, διότι δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε τα έγγραφα εργασίας και να μας δώσετε την άποψή σας εν το χρόνο, διότι και εμείς και οι σκιώδες εισηγητές επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή τους ακρογωνίους λίθους της έκθεσης αυτής και θα θέλαμε να ορίσουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε εδώ το Μάρτιο, τον Απρίλιο και να είμαστε ακόμα στην αρχή. Ε, να προσπαθήσουμε δηλαδή να αποφασίσουμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα ε, όλοι με μισείτε, αλλά αν πάτε σπίτι σας 6.30 για τις 8 θα με αγαπήσετε. Ο κύριος Ρούτσας, ευχαριστώ πολύ Σοφή, θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Καταρχάς θα ήθελα να αρχίσω κι εγώ ε, από την αγαπημένη μας προσέγγιση δέσμης ε, και την τηρούμε. Είναι γνωστό σε όλους, αφορά το μέθοδο εργασίας, το χρονοδιάγραμμα, αλλά και κάτι άλλο και θα ήθελα εδώ να παραθέσω αυτό που μας ζήτησε ο επόπτης προστασίας προσωπικών δεδομένων να κάνουμε ως νομοθέτες, ότι και ο κανονισμός και η οδηγία να έχουν τα ίδια βασικά στοιχεία και τις βασικές διατάξεις και να τεθούν σε ισχύ την ίδια ημέρα. Ε, αυτός είναι στόχος μας και θα τον τηρήσουμε. Η πολιτική πτυχή και πάλι ξέρουμε ποια είναι. Είναι απρόθυμα τα κράτη-μέλη για την οδηγία και επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι ακόμα η τρέχουσα Προεδρία δεν πιέζει για αυτό το θέμα όσο εμείς θα θέλαμε να ε, τη δούμε και γι' αυτό θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή ότι θα υποβάλουμε κοινοβουλευτική ερώτηση, προφορική δηλαδή ερώτηση και προς το Συμβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε να εγγραφεί στη μέση διάταξη της επόμενης συνόδου στο Στρασβούργο έτσι ώστε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα, να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί, αν θέλετε ακόμα και να ασκήσουμε κάποια πολιτική πίεση και είναι προφανές για όλους μας ότι όταν θα μας απαντήσουν στην Ολομέλεια και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα για το άμεσο μέλλον και τι θα κάνει το Κοινοβούλιο για την οδηγία. Δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Uh, Επί έχουμε το έγγραφο εργασίας, το οποίο έχει διανεμηθεί ήδη πριν την προηγούμενη διακοινοβουλευτική συνάντηση που είχαμε τη συνεδρίαση με συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων και κατά την άποψή μου αυτό ήταν πάρα πολύ επιτυχές ως εγχείρημα, ε, όσο και χρήσιμο αυτή η ανταλλαγή απόψεων και επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ ή να τονίσω ε, ορισμένα σημεία που αναφέρονται μεν στο έγγραφο εργασία, αλλά χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων και συζητήσεων. Πρώτον, και ξεκινώ από το θέμα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμοί, γραφεία κτλ. εκτός, ε, δεν εμπίπτουν μάλλον στο τομέα ε, εφαρμογή τη οδηγία, παρόλο που γίνεται ευρύτατη ανταλλαγή δεδομένων ε, σε τομεί επιβολή του νόμου και στο δικαστικό κλάδο. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και επίση στο ζήτημα του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση των ειδικών αυτών πράξεων στα πλαίσια τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία μία τριετία μετά τη θέση σε ισχύ τη οδηγία. Εγώ θεωρώ ότι πρακτικά αυτό σημαίνει τρία έτη συν Κάτι ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσουμε σε κοινά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστούν έξι χρόνια περίπου. Και για μας ένα τέτοιο χρονικό διάστημα και ένα τέτοιο χρονικό ορίζον είναι απαράδεκτος. Επίση, κάτι άλλο που πρέπει να συζητήθει περαιτέρω είναι το εξή. Έχουμε πολλές εξαιρέσεις στις αρχές που έχουμε θέσει. Δηλαδή μια βασική προστασία, μάλλον πώς να το πω, ε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αρχή είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και κάθε εξαίρεση θα πρέπει να τεκμηριώνεται, να δικαιολογείται και οι περιορισμοί να είναι εξαίρεση του κανόνα και να μην γίνουν ο κανόνας ο ίδιος. Άλλο θέμα είναι κάτι που έχει να κάνει και με τον κανονισμό. Ορισμένοι ορισμοί χρειάζονται περισσότερη διευκρίνηση ως στοιχεία δεδομένων ε, ε, διακράτηση, ε, ενημέρωση. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι τεχνική όρη ενδεχομένως. Θα πρέπει να συζητηθούν και να διευκρινιστούν ακόμα. Ε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης για μια σωστή αξιολόγηση ε, των αναγκών και ε, ένα είδος αναλογικότητας. Δεν υπάρχει και σαφής ορισμός του λεγόμενου profiling και ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο που αφορά ε, το καθεστώς που προτείνεται για μεταφορά ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες είναι ασαφής, είναι αδύνατος και δεν ε, περιλαμβάνει όλα τα εχέγγυα για να προστατεύονται τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα στοιχεία θα διαβιβάζονται. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει η αρχή να που είναι επιφορτισμένη ε, με την ε, προστασία και την ε, παρακολούθηση όλων αυτών δεν έχει ακόμα με σαφή τρόπο διατυπωμένο το πεδίο δράσης και λειτουργίας. Εμείς προτείνουμε και θα προτείνουμε τροπολογίες για να αυξηθεί η προστασία όπου χρειάζεται αντίστοιχη με τον κανονισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Λιμπάη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και πολύ σύντομα όπως ζητήσατε. Καταρχήν να πω ότι ορίζουν τα έγγραφα εργασία που παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σίγουρα θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, υποστηρίζουμε τις ε, προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε ότι υποστηρίζουμε την ιδέα να έχουμε μία κοινή γενική προσέγγιση στα τέλη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Συνειδητοποιούμε βέβαια ότι είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα θέλαμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, επί της ουσίας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά σημείων που τέθηκαν καταρχήν ε, από το Γιάνν Άλμπρεκτ για τις ε, θεμελιώδεις αρχές, για την κυριαρχή και για τον ε, αποσαφηνισμό του ορισμού. Συμφωνούμε να συνεργαστούμε, να εργαστούμε από κοινού και να βρούμε μια λύση αποσαφήνισης αυτών των σημείων. Για το θέμα που θέσατε επίσης, ε, για την ενδυνάμωση των ε, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, την απλούστευση και τη συγχώνευση διατάξεων, ευχαρίστως να εξετάσουμε το κείμενο στα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος, που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Έχουμε πει με σαφήνεια ότι Θέλουμε να ακούσουμε λύσεις που θα παρουσιαστούν για την μείωση, αν είναι δυνατόν για την ακόμη περαιτέρω μείωση του διοικητικού άχθους για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας και υπόψη πως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασία μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό για τις ε, μεγάλες εταιρείες ε, υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, εφαρμοστικές και τις κατεξουσιοδότηση πράξης, τις εκτελεστικές κατεξουσιοδότηση πράξης, με συγχωρείτε, καλωσορίζουμε τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν από τον εισηγητή. Έχουμε δηλώσει ότι ευχαρίστως να εξετάσουμε την πρόταση αυτή για τις κατεξουσιοδότηση πράξης, μία προς μία, βάσει των κριτήριων. αλλά έχοντας ε, και κατά νου το πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε και ευελιξία στον κανονισμό. Γιατί θα πρέπει να ακολουθεί και τις επιταγές της τεχνολογίας. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή για την ε, προσέγγιση της δέσμης μέτρων. Από την αρχή υποστηρίζαμε και φυσικά συμφωνήσαμε στο να εξετάζουμε και τον ορισμό τους ορισμούς, αναφερθήκατε σε κάποιους από αυτούς. Γενικά θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εισηγητές για να βελτιώσουμε τα κείμενα και να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που έχετε θέσει. Και πάλι έχοντας κατά νου ότι θέλουμε να αυξήσουμε τα δικαιώματα των ατόμων. Επίσης, θέλουμε να υπάρχει και μια διάσταση εσωτερικής αγοράς ε, στο θέμα της προστασίας των δεδομένων και θέλουμε να ενισχυθεί η διάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντρέο, εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο, αλλά και την ευκαιρία να ενημερώσουμε την Επιτροπή ε, για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το πακέτο των προσωπικών δεδομένων για την πρόταση κανονισμού και την πρόταση οδηγία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εργασίες που έχει κάνει η Κυπριακή Προεδρία από την τελευταία ενημέρωση που σας έχουμε κάνει εδώ στη LIBEC Committee μέχρι και τον επόμενο προγραμματισμό μας τον Δεκέμβριο στο Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ε, Υποθέσεων. Θα ξεκινήσω αναφέροντα ότι κατά τη διάρκεια του Οκτώβρη, στι 12 Οκτωβρίου, η Προεδρία διοργάνωσε την πρώτη ε, συνάντηση Friend of the Presidency, όπου συζητήθηκε ένα από τα οριζόντια θέματα που είχαμε θέσει στο άτυπο συμβούλιο ΔΕΗ e στη Λευκοσία, δηλαδή των κατεξουσιοδοτήσεων και εκτελεστικών πράξεων. Οι συζητήσει για το θέμα αυτό συνεχίστηκαν κατά τη διήμερη συνάντηση εμπειρογνωμόνων DAPIX Data Protection η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 του Οκτώβρη. Θα πρέπει να πούμε ότι στη διήμερη αυτή συνάντηση εξετάστηκε επίσης και η πρόταση κανονισμού, εξετάζοντας άθρο προς άρθρο τον κανονισμό, φτάνοντας μέχρι το άρθρο 39. Να υπογραμμίσουμε ότι οι συζητήσει κατά τη εξουσιοδότηση και εκτελεστικέ πράξει είχαν καταδείξει ότι υπήρχαν αρκετέ συγκλήσει μεταξύ των αντιπροσωπιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό των κατοξισοδοτήσεων πράξεων. Πολλέ από τι πράξει κρίθηκαν ομόφωνα υπερβολικέ ή αδικαιολόγητε σε σχέση με το περιεχόμενο των σχετικών άρθρων. Όσον αφορά τι εκτελεστικέ πράξει, για περιορισμένο αριθμό άρθρων, τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν την αναγκαιότητά του, αλλά και για την πλειοψηφία των άρθρων εκφράστηκαν ανησυχίε τόσο για την ανάγκη θέσπιση εφαρμοστικών πράξεων, όσο και με τη συμμόρφωση με τι διατάξει τη συνθήκη που παρέχουν στην Επιτροπή αυτή την εξουσία. Ταυτόχρονα θα πούμε ότι το θέμα των, προσωπικών δεδομένων, το πακέτο είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ΔΕΗ που είχε πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στι 26 Οκτωβρίου. Ο Υπουργό μα είχε ενημερώσει το Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά των φάκελων αυτών. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να πούμε ε, εδώ είναι ότι τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και πολιτικό επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο, η Επιτροπή εξέφρασε την ετοιμότητά τη όπω για το θέμα των κατεξουσιοδοτήσεων πράξεων κρατήσει μόνο τι απαραίτητε, δηλαδή ε, τη διαγραφή μέχρι και 40%. Αυτό όμω, όπω ανέφερε, θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια ενό επικοδομητικού διαλόγου με την εξέβρεση συμβιβαστικών ή και εναλλακτικών λύσεων. Περαιτέρω να αναφέρω ότι στο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση του θέματο αυτού είχαν εκφραστεί από ορισμένε αντιπροσωπείε οι ανησυχίε ω προ την κατά πόσο η πρόταση κανονισμό θα μπορούσε να ήταν οδηγία αντί κανονισμό. Να αναφέρω επίση ότι η Κυπριακή Προεδρία, στη βάση των συζητήσεων που έγιναν όσον αφορά το πρώτο οριζόντιο θέμα των κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, έχει ετοιμάσει έγγραφο το οποίο αναμένεται να αποσταλεί στα κράτη-μέλη με σκοπό να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 13 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης φίλη της Προεδρίας. Απότερος στόχος μας είναι όπως ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και το παρουσιάσουμε τόσο στην Κορεπέρ όσο και στο Συμβούλιο ΔΕΗ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα αναμένεται να ετοιμάσουμε δεύτερο έγγραφο σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουμε λάβει από τις αντιπροσωπείες για το δεύτερο οριζόντιο θέμα που αφορά το διοικητικό φόρτο. Το θέμα αυτό αναμένεται να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης DABIX Data Protection που θα γίνει στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Για το θέμα αυτό στοχεύουμε και πάλι να ετοιμάσουμε σχετικό έγγραφο όσον αφορά το διοικητικό φόρτο για να το παρουσιάσουμε επίσης τόσο στην Κοροϊπέρ όσο και στο Συμβούλιο του Δεκέμβρη. Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι η Προεδρία συνεχίζει να εργάζεται σκληρά και συλλογικά, όπως αυτό πράττει από την ανάληψη της Προεδρίας της για το φάκελο αυτό, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να δώσουμε στην ε, επόμενη Προεδρία χειροπιαστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Τέλο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλιόρα από τι νομικέ υπηρεσίε να παρουσιάσει, καθώ επίσης και του συναδέλφου που θέλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση να σηκώσουν τα καρτελάκια του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Είχα να απαντήσω σε ερωτήσεις όσον αφορά τον, το σχέδιο του κανονισμού σε δύο σημεία. Θα προσπαθήσω. Καταρχάς, τη σχέση ανάμεσα στο σχέδιο κανονισμού και την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές νομοθεσίες και έπειτα το ζήτημα των καταξουσιοδότηση πράξεων. Καταρχάς, η σχέση ανάμεσα στο σχέδιο του κανονισμού και στις εθνικές νομοθεσίες. Η σχέση αυτή πρέπει να αναλυθεί με φόντο τη νομική βάση, τους στόχους του προτινόμενου κανονισμού, αλλά και της επιλογής νομικού μέσου. Το σχέδιο κανονισμού βασίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διτό στόχο. Από τη μία την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και από την άλλη η απαλληφή των περιορισμών για την ελεύθερη ροή προσωπικών δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει τον κανονισμό στο νομικό μέσο και στην περίπτωση υιοθέτηση του κανονισμού αυτού το περιθώριο λιγμών για τι εθνικέ νομοθεσίε στον τομέα αυτό τη νομοθεσία θα γίνει μικρότερο από όσο είναι τώρα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να παρασχεθεί κάποιο χώρο για λιγμού ε, στι εθνικέ νομοθεσίε, ακόμα και σε περίπτωση κανονισμού, με τη μορφή εθνικών εφαρμοστικών μέτρων ή παρεκκλήσεων. Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να είναι σαφώς περιορισμένες και δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν στο σκοπό του νομοθετικού έργου στο σύνολό του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα εθνικά μέτρα δεν πρέπει να εμποδίσουν την ελεύθερη ροή των προσωπικών δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά την ερμηνεία της έκφρασης μέσα στα όρια του κανονισμού, που χρησιμοποιείται σε πολλές διατάξεις του σχέδιου κανονισμού, αυτή η διατύπωση σε γενικές γραμμές αποτρέπει τα κράτη-μέλη από το να υιοθετήσουν κανόνες οι οποίοι θα παρεκκλίνουν του κανονισμού. Επίσης, να διευκρινίσω ότι από την προοπτική των εθεμελιωδών δικαιωμάτων η διατύπωση αυτή είναι ουδέτερη, διότι μόνος της στόχος είναι να διασφαλίσει την συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τον κανονισμό. Τώρα, όσον αφορά μια πιθανή επιμήκυνση ε, συγκεκριμένων κανόνων που περιέχονται στο κεφάλαιο 9 της ε, πρότασης κανονισμού για, περιπτώσει για περιπτώσεις επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων, είναι δυνατή τροποποίηση. Ωστόσο, διατάξεις ε, αυτές πρέπει να παραμείνουν περιορισμένες στους τομείς όπου έχει κριθεί αναγκαίο και δικαιολογημένο. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να συμμορφώνονται με τον σκοπό της νομοθετικής πράξης. Δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερα εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση προσωπικών δεδομένων. Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε μια πιθανή τροποποίηση έτσι ώστε να εισαχθεί μια διάταξη που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πιο αυστηρούς εθνικούς κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά παρέκκληση από, το σχέδιο κανονισμού η τροποποίηση, έτσι όπως ε, διατυπώθηκε στο ερώτημα αυτό, δίνει στα κράτη-μέλη πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη και ευρία παρέκκληση, το οποίο θα αντίβαινε στην πρόταση και θα οδηγούσε σε περισσότερη νομική ασάφεια. Ω συμπέρασμα τώρα στο πρώτο μέρο, να υπογραμμίσω ότι είναι δυνατόν και πολλέ φορέ αναγκαίο να υπάρξει περιθώριο ελιγμών για τις εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, ε, οι εθνικοί κανόνες δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περισσότερους περιορισμούς στην ελευθερία ροή προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ορισμένες από τις ε, τροποποιήσεις που εξετάστηκαν, εάν υιοθετηθούν, θα αφήσουν στα κράτη-μέλη μια, πολύ ε, μεγάλη ένα πολύ μεγάλο περιθώριο ε, απόφαση όσον αφορά την εφαρμογή της ε, νομοθετικής πράξης αυτής. Η επιλογή του νομικού μέσου θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί και ίσως να αντικατασταθεί από οδηγία. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο μέρος της ε, νομικής γνωμοδότησης για τις καταξουσιοδότησης πράξης. Η νομική υπηρεσία ζητήθηκε να αξιολογήσει εάν κάποια από αυτές τις ε, κατεξουσιοδότες πράξεις θα αφορούν τα σημαντικά στοιχεία ε, του προτινόμενου κανονισμού. Τώρα, καταρχάς, σύμφωνα με την λομολογία του δικαστηρίου και σύμφωνα με τις συνθήκες, η ε, εξουσία να τροποποιηθούν ή να προσθεθούν μη αναγκαία στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης μπορεί να, να γίνει ε, με καταξουσιοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις αναγκαίες και στις μη αναγκαίες πτυχές μιας νομοθετικής πράξης. Και παρότι το δικαστήριο δεν έχει ερμηνεύσει την έννοια των ε, αναγκαίων στοιχείων σε σχέση με τις καταξουσιοδότηση πράξης, μπορούμε να πάρουμε διδάγματα από την ομολογία όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων πριν από την έναρξη ισχύς της θήκης της, της Λισαβόνας. Στην ομολογία το δικαστήριο ε, καθόρισε τα σημαντικά στοιχεία ως κανόνες οι οποίοι πρόθεση έχουν να δώσουν ένα συμπαγές σχήμα στις ε, βασικές κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις, αποφασίζοντας ότι τα αναγκαία στοιχεία είναι διατάξεις οι οποίες για να υιοθετηθούν απαιτούν πολιτικές επιλογές που υπόκεινται ε, στην ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ε, πούμε ότι οι διατάξεις που θα είναι μια μεγάλη εξέλιξη στην ευρωπαϊκή πολιτική μπορούν μόνο να ε, ληφθούν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πρόεδρος παρεμβαίνει. Κύριε Λογίλο, παρακαλώ ολοκληρώστε. Μάλιστα, θα συνοψίσω λοιπόν. Πιστεύω ότι ένας αριθμός των ε, προτινόμενων διατάξεων στο σχέδιο κανονισμού εξαρτάται από τον νομοθέτη και είναι στα χέρια του νομοθέτη να αποφασίσει ποιες από αυτές θα μπορούν να θεωρηθούν ως ε, πρόσθετα μη σημαντικά στοιχεία και τι θα θεωρηθεί στόχος σε αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πρόεδρος, παρακαλώ ολοκληρώστε. Μάλιστα, αυτά είχα να πω. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά την κοινή, το, το common understanding. Δεν είναι δεσμευτικές διατάξεις. Μπορείτε λοιπόν να λάβετε αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τέσσερις συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Βός πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, οφείλω να πω ή ε, θέλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία μας και καλό είναι έτσι όπως το έχουμε ρυθμίσει αυτό τον καιρό, ακόμα κι αν μπορεί ορισμένα να μπορούσαμε να τα είχαμε διεκπαιρεώσει ταχύτερα κτλ. Καλό είναι όμως που ε, ε, προχωρούμε με την ησυχία μας και παίρνουμε το χρόνο. Θέλω να επενέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ένα δελτίο τύπου της 16ης Οκτωβρίου και πραγματικά είναι ωραία ένδειξη και ειλικρίνειας και ευελιξίας. Και ε, υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε, αλλά υποθέτω ότι και εκεί θα δείξετε ευελιξία. Ε, τώρα, μεμονωμένα για τον κανονισμό. Βεβαίως έχουμε αρκετά θέματα που πρέπει να διευκρινίσουμε αφενός και που ε, αφορά ε, επιμέρους θέματα, ας πούμε ε, δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα στη λύθη ακόμα, να ξεχαστούν κάποια στοιχεία. Όλα αυτά δεν μπορώ να τα πω τώρα σε λεπτομέρειες. Είναι καλή αφετηρία πάντως για να βασιστούμε και να προχωρήσουμε. Και σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά την οδηγία, είναι σωστό ε, να κάνουμε αυτή την πρόταση. Ε, όλοι όμως θα επιθυμούσαμε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο το Συμβούλιο σε αυτά τα θέματα. Και επίσης ελπίζω το Συμβούλιο να αρχίσει να σκέφτεται όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις. Οπότε καλό θα ήταν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Το Κοινοβούλιο δηλώνει πρόθυμο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε λίγο το Συμβούλιο να δούμε. Ε, αν πατήσετε λίγο γκάζι θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς και τους δύο συγγητές. Νομίζω είναι πολύ καλή αυτή η εργασία και των δύο και τα έγγραφα εργασίας το καταδεικνύουν. Δείχνουν ότι έχετε συμπεριλάβει πολλά στοιχεία που προέκυψαν από τη συζήτηση, αλλά παραμένει η κριτική προς το Συμβούλιο. Βεβαίως θέλουμε την ίδια διαδικασία και στα δύο έγγραφα και βεβαίως ε, θα πρέπει να πιέσουμε χρονικά, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε ε, το διάστημα που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμα και προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου. Άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την προστασία δεδομένων δεν μπορούμε να τα λύσουμε αν δεν επέλθει σαφήνεια για αυτά τα δύο πακέτα αν θέλετε να συζητήσουμε τα PNR και άλλα θέματα επιβατών και καθημερινά, αλλά αν δεν έχουμε ρυθμίσει ξεκάθαρα τα θέματα αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτό το τομέα, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και τίποτα άλλο, ούτε για τα δεδομένα των επιβατών, ούτε να δεσμευτούμε για τίποτα άλλο. Ήθελα να το πω αυτό, να ακουστεί. Τα δικά μας προβλήματα έδειξαν τους τελευταίους μήνες ότι είναι τα θέματα το πεδίο εφαρμογής, το είπαν και οι συγητές ε, ότι μας αφήνει μια πικρία το γεγονός ότι εξαιρούν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Ε, πώς γίνεται η προστασία των δεδομένων στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εγκριθούν διάφορες διατάξεις. Τι θα πει αυτό, δεν μας ικανοποιεί. Και τα διαφορετικά πρότυπα. Στο ένα πακέτο έχουν έτσι και στο άλλο αλλιώς. Ε, αυτές τις διαφορές τις βλέπουμε ακριβώς εκεί. Και εκεί που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή τα δικαιώματα ε, των ενδιαφερομένων που είναι πάρα πολύ χαλαρή η ρύθμιση και μιλάω για την οδηγία κυρίως. Αν θέλετε να τα δούμε άρθρο προς άρθρο, αλλά ας το αφήσουμε καλύτερα τώρα. Ε, άμα το δει κανεί έτσι πιο προσεκτικά το καταλαβαίνει αμέσως. Ε, το όλο θέμα των τρίτων χωρών. Εγώ έχω ένα πρόβλημα αρχής. Δηλαδή, τι θα πει με την αναλογικότητα, δηλαδή όταν υπάρχει δεδομένη προστασία ε, ή η κατάλληλη προστασία και αυτό πώς ορίζεται. Ε. Και αυτό το θέμα με τις κατεξουσιοδότηση πράξης πραγματικά με συναρπάζει. Καλό είναι και θέλω να μου εξηγήσετε πώς ορίζεται ο ρόλος ουσιώδες, essential. Γιατί Τελειώνεται, λέει η Πρόεδρος. Ναι, ωραία. Χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση αυτός ο όρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Uh, thank you, Chairman. I have already comment. Ευχαριστώ. Ήδη έχω σχολιάσει επανειλημμένο uh, το θέμα τη αποθήκευση των δεδομένων και ευχαριστώ τι ευκαιρίε uh, που έχουμε να συνεργαστούμε καλά για να έχουμε ασφαλή δικαίου. Πρέπει να διευκολύνουμε την εφαρμογή. Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Ένα που αφορά τα παιδιά και ένα που αφορά την ισορροπία μεταξύ της δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα και την προστασία των δεδομένων. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα κανόνων ε, που θα είναι ευνόητοι σε σχέση με τη συγκατάθεση και υπάρχουν, ε, αν και υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για τα παιδιά για το θέμα της συγκατάθεσης, όμως δεν υπάρχει ε, ένα σαφής κανόνας για το τι γίνεται με τα παιδιά πάνω από τα 13 έτη. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη διάταξη για τα παιδιά που είναι άνω των 13 ετών, κάπου παρ' το να ε, ζητείτε η ημερομηνία γέννηση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωση. Να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουν τα παιδιά περί τίνο πρόκειται. Για κατόπιν υπάρχει μια ε, αναφορά στη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. ρωτήσουμε πώ μπορούμε να την ενδυναμώσουμε. Γιατί προστατεύοντας τα δεδομένα, δεν θα έπρεπε να υποσκάπτουμε την πολύ σημαντική έννοια της πλήρους πρόσβασης στα δημοσία έγγραφα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ήσασταν πολύ σύντομοι. Κάποιο άλλο συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο. Όχι, τότε και εγώ σκιώδης ε, θα πάρω το λόγο, μήπως μπορείς να βάλεις ε, το χρόνο να τρέχει και θα με σταματήσω. Υποστηρίζω καταρχήν την προσέγγιση της δέσμης μέτρων, ε, αν και θα προτιμούσα να έχουμε ένα και μόνο μέσο, τώρα έχουμε δύο. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, η οδηγία να αποδυναμωθεί, να είναι ένα πολύ πιο δύναμο μέσα από το κανονισμό. Ξέρω ότι το Συμβούλιο όχι μόνο καθυστερεί το έργο της οδηγίας, αλλά υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη τα οποία ζητούν ε, να υπάρχουν μέσα στην οδηγία ε, κάποια θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας και να μην μπουν στον κανονισμό. Έτσι λοιπόν ε, τελικά θα έχουμε τις δημόσιες αρχές να κάνουν ό,τι θέλουν με τα δεδομένα όπως ε, κάνουν και σήμερα αλλά κατόπιν θα το κάνουν νόμιμα. Ε, συμφωνώ με την κυρία Έγνιστε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω πρόταση για την δικαστική και αστυνομική συνεργασία που μας ζητείτε να υιοθετήσουμε εμείς, μας ζητείτε από το Συμβούλιο να υιοθετήσουμε, μπορούμε να την υποστηρίξουμε μόνο αν το Συμβούλιο υιοθετήσει την οδηγία εγώ δεν θα ψηφίσω οτιδήποτε παρά μόνο αν είναι ισορροπημένο. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Και τέλος, για να αναφερθώ συγκεκριμένα στον κανονισμό, Νομίζω ότι ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να είναι πιο ευέλικτα. Θα έπρεπε να επιλέξουμε μια προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στον ε, κίνδυνο παρά στον κανόνα. Και αυτό θα ε, εξυπηρετήσει το συμφέρον και των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Μα έμειναν και 8 δευτερόλεπτα, λέει ο μιλήτρια. Κάποιο άλλο συνάδελφο θέλει το λόγο. Όχι, τότε να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει σε συντομία στα θέματα που τέθηκαν και θα ξαναδώσουμε το λόγο στους συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, από την παρέμβασή σας εννοώ ότι υπάρχει πολλή υποστήριξη για όσα υπάρχουν επιτάπητος και φυσικά τέθηκαν διάφορα ζητήματα και το κύριο μήνυμά μου σήμερα είναι να πω ότι είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε πολύ επικοδομητικά με το συνομοθέτη. Στο προηγούμενο συμβούλιο συνομίλησα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και σήμερα θέλω να σας διαβιβάσω το δύο μήνυμα. Υπάρχουν ε, πολλές επικοδομητικές προτάσεις ε, που ακούγονται και πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουμε δώσει το μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε ε, στα πλαίσια κατεψουδότησης πράξεων, πρέπει να το σχάρει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρούμε λύσεις πολύ σύντομα Βάση κριτηρίων. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα επί των οποίων νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια ταχύτατη λύση. Για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τώρα που τέθηκαν, πρέπει να το για τα παιδιά Αναφερθήκε σε αυτό κύριε Κορέτσα Μπίλτ. Ναι, έχουμε βάλει αυτό το ηλικία 13 ε, ετών για τα παιδιά και να σας πω ότι ευχαριστώ ε, να διερευνήσουμε καλές δυνατότητες. Απλά θέλω να σας επισημάνω ότι από τεχνικής άποψης είναι πολύπλοκο το θέμα να το επιλύσουμε. Όμως από τις αρχές ε, φυσικά ευχαριστώ να το εξετάσουμε όπως ευχαριστώ και να εξετάσουμε το θέμα της ε, πλήρους πρόσβασης στα δημοσία έγγραφα. Και για όσα είπατε, Πρόεδρε, για την τάση που υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη να προτιμούν να, να μπουν στην οδηγία όλα έχουν να κάνουν με τις δημόσιες αρχές, το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύση και ευελιξία εντός του κανονισμού για να απελευθούν τα προβλήματα που τέθηκαν σε ό,τι αφορά την προσέγγιση βάση κινδύνου που αναφέρατε. Είμαστε υπέρ ε, του να αυξήσουμε την προσέγγιση αυτή βάση κινδύνου στο κείμενο του κανονισμού, όμως ε, πρέπει να είναι απλό το κείμενο. Και η προσέγγιση βάση κινδύνου θα μας ε, εξαναγκάσει να εξετάσουμε τους κινδύνους που μπορεί να ενέχονται για κάθε άτομο, όμως στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, θα είναι δύσκολο, γιατί στην περίπτωση αυτών ο κίνδυνος είναι περιορισμένος συνήθως. Επίσης έχουμε προτείνει με τέτοια προσέγγιση στον κανονισμό και είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε και πρόσθετα στοιχεία για να ενδυναμώσουμε αυτή την προσέγγιση βάση κινδύνου για το χρονοδιάγραμμα γενικά. Είπατε ότι το υποστηρίζετε ένθερμα. Να σας επισημάνω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία πολύ φιλόδοξα ως προς το χρονοδιάγραμμα και πάλι να σας πω ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψω στην ερώτηση τη κυρία Κορέτσα Μπίλτ για τη σχέση ανάμεσα στην προστασία δεδομένων και την πρόσφατα στα έγγραφα. Είστε ευχαριστημένοι από την απάντηση. Μάλιστα. Θα ήθελε το Συμβούλιο, η Προεδρία να απαντήσει. Εν όχι τότε επιστρέφουμε στους συζητητές. Κύριε Δρούτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Σόφη. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Απλά να πω ότι είμαι ευγνώμων που σας έχω στο πλευρό μου για την προσέγγιση δέσμης και, αλλά και για το ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα που θα στείλουμε. Είναι πολύ καλό να υπάρχει μία φωνή δυνατή. Να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά την Επιτροπή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θα ήθελα ξανά να τονίσω το ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετική σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά γι' αυτό. Ιδιαίτερα για το ότι συμμεριζόμαστε, ε, την ίδια προσέγγιση για, την, ε, για το μέλλον της οδηγίας και επίσης να διευκρινίσω ότι όλα τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί δεν είναι κριτική. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία επίσημα να τονίσει την θέση με τις προφορικές ερωτήσεις που είχε και στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι σύντομος. Είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτήν την οδηγία. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε ότι θέλουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των ε, δεδομένων και απαιτούμε να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την προστασία δεδομένων σε αυτόν τον τομέα. Αυτό λοιπόν απαιτούμε και εργαζόμαστε γι' αυτό σκληρά, συνεργαζόμαστε. Θα υποβάλουμε πρόταση από πλευράς μας και είμαστε ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν πιστεύω πως πρέπει να συζητήσουμε για πιθανότητες ε, την παρούσα στιγμή, αλλά να παρουσιάσουμε αποτελέσματα για αυτήν την οδηγία. Έπειτα, φυσικά, είναι και αναγκαίο, γιατί υπάρχουν προτάσεις όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας, ε, για τις οποίες μας έχει ζητηθεί να τις εξετάσουμε και άλλοι φάκελοι στον τομέα αστυνομική συνεργασίας, όπου η δική μου τουλάχιστον ομάδα πιστεύει ότι τα ελάχιστα πρότυπα όπως θα ενσωματωθούν από εμάς στην οδηγία για την προστασία δεδομένων, είναι αναγκαίο να υπάρχουν εκεί προτού υιοθετήσουμε μέτρα για ανταλλαγή πληροφοριών ε, όσον αφορά τις αρχές επιβολής νόμου. Αυτά από εμάς για αυτό. Τώρα επιστρέφοντας στον κανονισμό, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που συνείσφεραν, ιδιαίτερα κυρία Κορότσα Μπίλτ, εάν έχετε κάποια πρόταση για το ζήτημα των παιδιών, κάτι το οποίο και εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, αλλά και για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, θα ήθελα πάρα πολύ να τη συμπεριλάβω στην οδηγία από την αρχή διότι έχω την εντύπωση ότι η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα σε πολλά κράτη-μέλη είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και πρέπει να υπάρξει μια σαφής ε, αναφορά στον κανονισμό για να μπορέσουν έτσι και οι αρχές προστασίας δεδομένων να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα μαζί. Και όσον αφορά τώρα την προστασία δεδομένων των παιδιών, Πιστεύω πως ιδιαίτερα για τα παιδιά πάνω από 13 χρονών θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά όσον αφορά το profiling. Και επίσης αναφορά ιδιαίτερα στα παιδιά όσον αφορά την συνένεση μετά από πληροφόρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ η Πρόεδρος προβλέπεται η κατάθεση των σχεδίων έκθεσης για τη συνεδρίασή μας 17 και 18 Δεκεμβρίου της Επιτροπής μας ε, χριστουγεννιάτικα δώρα. Λοιπόν, τώρα που σας πίεσα όλους να είμαστε επιθαρχημένοι, τελειώσαμε 8 λεπτά νωρίτερα. Και σας ζητώ συγγνώμη. Ε, αύριο μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση 8 λεπτή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ραντεβού αύριο.